σε αυτός θα αναφέρεται και θα ισχύσει για την ανανέωση των μελλοντικών εντολών στα πλαίσια της κοινοβουλευτική δραστηριότητας. Κύριε Άοντι, τις παρατηρήσεις σας τις άκουσα προσεκτικά εκ προημίου αναφέρεσαι σε μια αναδρομική εφαρμογή. Ωστόσο αυτό δεν επιτρέπεται από τον κανονισμό μας. Παρακαλώ να δείξετε κατανόηση γι' αυτό. Ότι πρέπει να κάνουμε αυτό το οποίο προβλέπει η Επιτροπή Κανονισμού και το οποίο η οποία Επιτροπή Κανονισμού σύμφωνα με την επιθυμία της Ολομέλειας μας υπέβαλε την πρόταση. Η ερμηνεία του άρθρου 191 είναι σαφής. Ζητώ κατανόηση για το ότι δεν μπορώ να αλλάξω αυτό αναδρομικά. Στην πολιτική όπως και στην ανθρώπινη ζωή δυστυχώς συμβαίνει αυτό. Αναδρομικά τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει εκ των υστέρων. Και αυτό πρέπει να το α, δεχτεί κανείς. Λυπούμε γι' αυτό. Και περνάμε στη συνέχεια στο πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης της σημερινής συνεδρίασης. Είναι η κοινή συζήτηση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τους ίδιους πόρους. Θα ακούσουμε τα όσα έχουν να μας πούν οι εισηγητές για την προσωρινή έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον πολιετή σχεδιασμό 2014-2020 από πλευρά του Ευρωκοινοβουλίου. Προτού δώσω τον λόγο στους εισηγητές, μια σύντομη παρατήρηση από πλευράς μου. Κατά τα, τους τελευταίους 6-7 μήνες είχα την ευκαιρία με την όπως την αποκαλούμε ομάδα επαφών που έχει αναλάβει τις διαπραγματεύσεις για εξ του Κοινοβουλίου με τα άλλα θεσμικά όργανα, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, προετοιμάστηκαν όλα αυτά και υπήρξε στενή συνεργασία. Και έτσι και σε σχέση με την ιδιότητά μου θα ήθελα εδώ στην Ολομέλεια να αναφέρω την εξαιρετική ποιότητα αυτής της ομάδας επαφών. Έχουμε τους διαπραγματευτές μας σε αυτή την ομάδα, τον κύριο Λαμαζούρ, τον κύριο Μπέγκε, τον κύριο Κάλφιν και τον κύριο Ντεχάνε, που εξ ονόματος του Ευρωκοινοβουλίου διεξάγουν τις γενικές διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Και στην ίδια την ομάδα συμμετέχουν και οι συντονίστρες και συντονιστές καθώς επίσης και το Προεδρείο της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Πρέπει να σας ομολογήσω και να σας πω κυρίες και κύριοι ότι είναι μια πραγματικά εξαιρετικά ικανή και ομάδα και πολύ ε, φιλική συνεργασία η οποία διασφαλίζεται που εκπροσωπεί το Ευρωκοινοβούλιο με τέτοιο τρόπο αναβαθμισμένα ποιοτικά που σπάνια το έχει ζήσει κανείς αυτό, εγώ τουλάχιστον και χωρίς να θέλω να μειώσω τις επιδόσεις των άλλων θεσμικών οργάνων μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για την ποιότητα εργασίας που έχουν ως επίδοση αυτές οι κυρίες και αυτοί οι κύριοι. Θα ήθελα εδώ να το αναφέρω αυτό και να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για αυτό το έργο τους. Θερμά καλοχαιρετίζω στη συζήτησή μας τον κύριο Μαυρογιάννη και τον κύριο Τσεφτιοβιτς και τον κύριο Λεβαντόφσκι, Λεβαντόφσκι που αναγκαία πρέπει να παρίστανται σήμερα το πρωί. Καλώς ήρθατε θερμά, κυρίες και κύριοι, στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου. Πρώτος θα λάβει τον λόγο ο εισηγητής για την προσωρινή έκθεση, ο κύριος Μπέγκε. Με τη σειρά θα τα πάρουμε, μετά ο κύριος Κάλφιν. Παρακαλώ κύριε Μπέγκε, έχετε τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να πω στην διαπραγματευτική ομάδα ανήκει και η κυρία Γένσεν, συνάδελφος από την Άλντε, την ομάδα των φιλελευθέρων. Να το αναφέρω αυτό. Ζητώ συγγνώμη, λέει ο πρόεδρο. Δεν είχα καμιά κακή πρόθεση να αγνοήσω, αλλά ήταν σοβαρό ολίσθημα αυτό. Φυσικά ισχύουν οι έπαινοι και οι ευχαριστίε και για την κυρία Γένσεν, για την ομάδα επαφών. Σα ευχαριστώ που το επανορθώσατε αυτό, κύριε Μπέγκε, και με τόσο φιλικό τρόπο. Μάλιστα, οι αρμόδιοι για τα δημοσιονομικά βλέπετε κύριε Πρόεδρε πως έχουν κάθε μικρολεπτομέρεια. Και γι' αυτό θα ήθελα να πω ότι το χαιρετίζω θερμά πόσο έντονα εσείς ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καταβάλατε προσπάθειες για τον εκδημοκρατισμό της δημοσιονομικής μας πολιτικής. Πέρα από κάποιες ε, διαφορές που υπάρχουν σε σχέση με τη συνέντευξή σας που δώσατε την ε, ε, Κυριακή το βράδυ. Ο κύριος Κάλφιν και εγώ υποβάλλουμε μια κοινή έκθεση που στο τέλος θα συνεισφέρει, όπως είναι η πρόθεσή μας, η διαδικασία έγκρισης για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο να επιταχυνθεί και να διευκολυνθεί. Το κάνουμε αυτό με βάση της εργασίας που έγινε ήδη στο παρελθόν της ε, ειδική Επιτροπής, της Επιτροπής ε, ΣΟΥΡ, της Ιούτα Χάουγκ, του Σαλβαδόρ Γκαρίγα. Θέλω να ευχαριστήσω ρητά και την προηγούμενη και τη σημερινή Προεδρία διότι βρισκόμαστε σε ένα είδους πιλωτικό σχέδιο, πιλωτικό πρόγραμμα πριν από την συνάντηση ε, του, Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και για τα όλα όσα συζητούνται υπό το ε, box το οποίο πρόκειται και έχουν προσκληθεί και οι εκπρόσωποι του Ευρωκοινοβουλίου στην άτυπη συνάντηση του ε, Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει η αμοιβαία εμπιστοσύνη να προαχθεί, να μπορούμε να εργαζόμαστε με ένα πιο έντονο τρόπο και να μην υπάρχουν προκαταλήψεις. Αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα, αυτή η μέθοδος εργασίας φυσικά όμως δεν δεν διασφαλίζει το τελικό αποτέλεσμα, την τελική έκβαση. Κατά τα άλλα, η ανάλυση μας ασχολείται περισσότερο από ότι με ένα μαγικό αριθμό. Εργαστήκαμε σε σχέση με τα θέματα παγκοσμιοποίησης με βάση τα μέχρι σήμερα πολιετή προγράμματα είδαμε πώς έχουν οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πώς πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Για μας φυσικά πρόκειται για ποσά, για λογικά, ορθά Πρόκειται για θέματα ουσίας, για μια ευρύτερη ελαστικότητα για την δημοσιονομική διαδικασία, για ίδιους πόρους που πραγματικά πρέπει να αξίζουν το όνομα, την ονομασία ίδιοι πόροι. Και σε αυτή τη συγκυρία πρόκειται ιδιαίτερα για τον ενιαίο χαρακτήρα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, όπως και από τη συνθήκη ε, χαρακτηριστικά και σαφώς καθορίζεται. Και υπάρχουν κάποιοι οποίοι μιλούν για ένα μαγικό αριθμό και λένε ότι στην πολιτική συνοχή ή στην, τη γεωργία όλα πρέπει να παραμείνουν ως έχουν και δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Αυτό όμως κυρίε και κύριοι δεν είναι συνεισφορά για, μια, για την ανάπτυξη σε μια δύσκολη συγκυρία. Αν τα κράτη-μέλη δεν είναι πρόθυμα να διαθέσουν κονδύλια επαρκή στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, τότε παρακαλώ να μας πούν επαρκώς ποιες πολιτικές προτεραιότητες αποφάσισαν τα ίδια γιατί δεν είναι δυνατό να αγνοηθούν αυτά τα γεγονότα. Δεν μπορεί να γίνεται επιτυχίες όπως ο Έρασμος με 2,5 εκατομμύρια φοιτητών να υφίστανται περικοπές επειδή κάποια άλλα πράγματα θέλει κάποιος να διατηρήσει στην πολιτική συνοχή ή αλλού. Δεν γίνεται να πούμε 3% για την έρευνα και ανάπτυξη και θα περικόψουμε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον χρονορίζοντα 2020. Δεν γίνεται να λέμε η Ευρώπη πρέπει να προσανατολίζεται σε ένα νέο ρόλο στην ε, πολιτική, την εξωτερική και την πολιτική ανάπτυξης και να έχουμε το 0,7% να μην τηρούμε καν το 0,7% του ΑΕΠ για την πολιτική ανάπτυξη. Αυτό δεν είναι αξιοπιστία φυσικά. Και χρειαζόμαστε Πάντα λαμβάνοντα υπόψη την εξυγίανση των δημοσιονομικών των κρατών μελών, κέντρο βάρου που θα δώσουμε στο better spending, στην καλύτερη διάθεση των δαπανών, των κονδυλίων. Ιδιαίτερη δουλειά για το διοικητικό τομέα και τα προγράμματα διαχείρισης πρέπει να γίνει και γίνεται για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Λέμε ταυτόχρονα ότι φυσικά τέτοια προγράμματα όπως συνδέοντας την Ευρώπη, Connecting Europe και η διαβίου ε, εκπαίδευση δεν μπορούν να αγνοηθούν και να τεθούν στο περιθώριο. Και λέμε το ότι σε σχέση με το θέμα του τι επικουρικά θα ρυθμίζεται και που υπάρχει ένα επικοδόμημα, ε, όλα αυτά πρέπει να συνεξεταστούν. Και σε σχέση με τα κράτη-μέλη που έχουν ε, εκατοντάδες πρεσβείες, προξενία και μυριάδες ατόμων που ασχολούνται εκεί και με τεράστιο προϋπολογισμό. Αυτό είναι 15% περισσότερο από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Υπηρεσίας ε, για το 2012. Και αυτό ανήκει ως στοιχείο στην συνολικότερη εικόνα της αλήθειας και της αντικειμενικότητας κυρίες και κύριοι. Και όταν λέμε ότι καταρχήν Θέλουμε να έχουμε ποσά, κονδύλια, με βάση τις αναλύσεις και τις νέες προκλήσεις που μας θέτει ενώπιόν μας η συνθήκη της Λισαβόνας και που ξεπερνούν τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όλα αυτά βασίζονται σε αυτή την ανάλυση ακριβώς. Αλλά κυρίες και κύριοι πρέπει να το γνωρίζει αυτό το Συμβούλιο. Σε περίπτωση μη συμφωνίας ε, δεν θα διαλυθούν τα πάντα. Θα παραμείνουν τα ανώτατα ανώφλια μέχρι ότου υπάρξει τελική λύση του προβλήματος. Αλλά ακριβώς η προσφορά που κάνουμε, η εξισορρόπηση μεταξύ των αναγκαίων ορθών κονδυλίων και όσο πιο δύσκολα είναι το, τα κονδύλια τόσο μεγαλύτερη ελαστικότητα χρειαζόμαστε. Να πούμε σαφώς, χρειαζόμαστε ίδιους πόρους όπως ο Ζαν Λουκ Ντεάνα και η κυρία Γένσεν το συμπεριέλαβαν στην έκθεσή μας. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν υποβάλλει μια ενδιαφέρουσα πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τον φόρο χρηματοοικονομικών συναλλαγών και μια μείωση των εθνικών εισφορών και τα συναφή. Και σε αυτό ανήκει επίσης όταν μιλάμε για ένα ε, ευρωπαϊκό μέσο διευκόλυνσης. Έχω έξι λεπτά. Το ευρώ είναι η περίπτωση η κανονική και ομαλή και όχι η εξαίρεση. Εδώ επιμένουμε και εμένουμε στον ενιαίο και ολοκληρωμένο χαρακτήρα του προϋπολογισμού ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να διασφαλίσει το μέλλον της. Και όταν το τέλος χρηματοοικονομικών ε, ε, συναλλαγών για την ε, διευκόλυνση για το μέσο του ευρώ, όποιος δεν θέλει να το κάνει αυτό δεν μπορώ να κατανοήσω αυτή τη λογική. Αυτό τα θεωρούμε ως στοιχεία του πυρήνα για αυτό το περιεχόμενο. Να είμαστε σε θέση γοργά να διαπραγματευτούμε και ταχαίως να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα. Αλλά όχι έναντι ουδήποτε αντιτίμου. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Μπέργκερ. Θα ήθελα στην ομάδα σας να πείτε πόσο γενναιόδωρα αντιμετώπισα τον χρόνο κατά τον οποίο είσαστε αγορητής. Ο κύριος Κάλφιν παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ, να πω ότι η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το πολιετές ε, πλαίσιο είναι κάτι το οποίο έχει ήδη συζητηθεί μέχρι τώρα. Ρόλος της έκθεσης αυτής είναι ξεκάθαρος. Να ενημερώσει το Συμβούλιο που θα συνεδριάσει στο τέλος ε, του μηνός, πριν συνεδριάσει, και θα εκφράσει ξεκάθαρα τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το επόμενο χρηματοοικονομικό πλαίσιο. Η συνθήκη λέγει ότι μπορεί να καταλήξει σε μία θέση το Συμβούλιο εφόσον έχει εκφραστεί η άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εκ των προτέρων λοιπόν προσπαθούμε να ενημερώσουμε για τις θέσεις του Κοινοβουλίου και γι' αυτό προετοιμάσαμε την έκθεση αυτή η οποία ελπίζουμε να γίνει δεκτή με μεγάλη πλειοψηφία σήμερα. Η έκθεση αυτή είναι ξεκάθαρη και στηρίζεται θα έλεγα από όλε τις πλευρές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά από συζητήσεις που ε, κράτησαν δύο χρόνια. Έχουμε συζητήσει το θέμα σε διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές, έχουμε υιοθετήσει πολλές επιμέρους εκθέσεις και έχουμε δείξει ότι υπάρχει μια ενότητα η οποία διαπερνά τις διαφορές ανάμεσα στις ε, πολιτικές ομάδες και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το ε, πλαίσιο αυτό είναι ένα μέσο, δεν είναι ένα απλό ε, θα έλεγα λογιστικό πλαίσιο αλλά είναι ένα πολιτικό μέσο το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας. νομίζω ότι και ο κύριος Λεβαντόφσκι, ο επίτροπος Λεβαντόφσκι και η Προεδρία έχουν, η Κυπριακή Προεδρία έχουν κάνει ό,τι μπορούν έτσι ώστε να εντάξουν το Κοινοβούλιο στη διαδικασία. Θέλω να τους ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω και εσάς κύριε Πρόεδρε του Κοινοβουλίου και όλους τους συναδέλφους που συνεργάστηκαν γιατί όπως είπα το θέμα αυτό μας ενώνει εδώ στο Κοινοβούλιο και αυτό καθιστά την απόφασή μας ισχυροτέρα. Τέσσερα σημεία σχετικά με τον προϋπολογισμό. Πρώτον, το μέγεθος του προϋπολογισμού. Ξεκινώντας θα ήθελα να πω ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ανεπαρκής για να χρηματοδοτηθούν όλες οι αποστολές τις οποίες έχει αποφασίσει η Ένωση και αυτό είναι σαφές. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο σχεδιασμός του επόμενου χρηματοοικονομικού πλαισίου γίνεται σε ένα πολύ ε, δύσκολο πλαίσιο. Έχουμε τα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη δυσκολία να τα ξεπεράσουμε και την ανάγκη για δημοσιονομική πειθαρχία και λιτότητα και περικοπές σε επίπεδο χωρών. Καταρχάς, ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν δημιουργεί ελλείμματα. Δηλαδή οι προσπάθειες των κρατών να, να τακτοποιήσουν τα δημοσιονομικά τους επειδή ξόδευαν πολύ περισσότερο τα τελευταία χρόνια δεν ισχύουν για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Δεύτερον, ο προϋπολογισμός ο ευρωπαϊκός είναι επενδυτικός προϋπολογισμός. Κάνει αυτά τα οποία δεν μπορούν να κάνουν οι εθνικοί προϋπολογισμοί λόγω ακριβώς των περιορισμών και περικοπών. Τρίτον, ο προϋπολογισμός αυτός έχει νόημα λόγω ακριβώς της μόχλευσης και των επιπλέον ποσών που προσελκύει για ε, επενδύσεις. Το 90% του προϋπολογισμού πηγαίνει πίσω στις χώρες και ε, προσελκύει πολύ περισσότερα χρήματα πολλές φορές. Λοιπόν, ε, μειώσεις στον κοινοτικό προϋπολογισμό σημαίνει επιπλέον μειώσεις για τη γεωργική πολιτική, τις περιφερειακές πολιτικές, την κοινωνική πολιτική κτλ. Πάρα πολύ συχνά ακούμε από τους εκπροσώπους των κυβερνήσεων ότι οι πολίτες δεν δέχονται έναν μεγαλύτερο κοινοτικό προϋπολογισμό. Θα πρέπει να τους πούμε εδώ ότι εμείς έχουμε ε, σωστή επαφή με τους πολίτες και ακριβώς οι πολίτες περιμένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους ηγέτες τους να συνεργαστούν και να προτείνουν ένα μηχανισμό εξόδου από την οικονομική κρίση, δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και ανάπτυξης χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ας μην φέρουμε σε αντίθεση λοιπόν το ευρωπαϊκό επίπεδο και τον ευρωπαϊκό προπολογισμό με τους εθνικούς αντίστοιχους. Αν κάποιες κυβερνήσεις επανέρχονται σε κάποια υπαρξιακά ερωτηματικά του είδους θέλουμε περισσότερη Ευρώπη, μπορούμε να δουλέψουμε στην Ευρώπη τότε αν θέλετε να μπούμε στη συζήτηση αυτή εφόσον βέβαια δεν είναι σαφές το θέμα για κάποιες από τις κυβερνήσεις. Ο κ. Μπέγκε αναφέρθηκε επίση στην ευελιξία του προπολογισμού. Η ευελιξία σε ένα περιορισμένο προπολογισμό δεν είναι κάτι το τεχνικό, το λογιστικό. Είναι η ικανότητα του να κατανείμει τι πιστώσει με τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο. Να τώρα κάποιες προτεραιότητες από το περιεχόμενο. Έχουμε τις λεγόμενες παραδοσιακές πολιτικές, αλλά για τα επόμενα 7 χρόνια θα πρέπει ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός να κινητοποιήσει την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι ο στόχος ενός προϋπολογισμού ευρωπαϊκού. Είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε όλες τις ιδέες σχετικά με μια καλύτερη κατανομή των δαπανών και πιο αποτελεσματική κατανομή των δαπανών, αλλά απαιτείται να υπάρξει ο προπολογισμό αυτός για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ειδικά του νέους. Και πολλές φορές και ο πρόεδρος της Επιτροπής έχει αναφερθεί στο θέμα της ανεργία των νέων εδώ. Και μια τελική ε, παρατήρηση για τις διαδικασίες. Θα ήθελα να πω εδώ κάτι το οποίο έχουμε επανειλημμένα τονίσει στις Προεδρίες, ότι το MFF ακολουθεί δύο διαδικασίες. Τη διαδικασία συνένεσης για τα θέματα τα οικονομικά και την ε, συναπόφαση για 70 ε, περίπου νομικές βάσεις. Εμείς δεν θέλουμε το Συμβούλιο να πάρει αποφάσεις για τις διαδικασίες τις οποίες εμπλέκεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς θέλουμε να διαπραγματευτούμε με τα κράτη-μέλη και με το Συμβούλιο σε όλα τα θέματα που άπτονται του προπολογισμού. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κάλφιν. Για σας ισχύει το ίδιο. Αυτό το οποίο είπα πιο πριν στον κύριο Μπέγκε για τη γενεοδορία στον χρόνο. Τον λόγο θα έχει τώρα ο πρόεδρος της, πολιτική, της Επιτροπής Προϋπολογισμών, συνάδελφος Λαμασού. Ευχαριστώ πολύ. Είστε, είστε πολύ γενναιόδωρος για αυτά που μας είπατε και για τον τρόπο που στηρίξατε τη δουλειά που κάνουμε στην ομάδα μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριοι επίτροποι, θα ήθελα να επιμείνω σε δύο σημεία τα οποία είναι κομβικά για το Κοινοβούλιο. Πρώτα απ' όλα, δεν θα συμφωνήσουμε για το ΠΔΠ εάν δεν υπάρξει μια πολιτική συμφωνία για την ε, αναδιάρθρωση των πόρων. Θα πρέπει δηλαδή να ξαναδούμε ποιοι είναι οι διορθωτικοί μηχανισμοί, ποιοι είναι οι νέοι ήδη οι πόροι και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα θέση σε ισχύ αυτών πριν συμφωνήσουμε. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αναμονή. Κανείς, δημοκρατικός, κανείς δημοκράτης δεν μπορεί να στηρίξει το σύστημα χρηματοδότησης του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Ξέρετε πως τα ε, rebates που έχουν κάποια κράτη ε, έχουν ήδη ε, καταπέσει δικαστικά και ξέρετε πως η διαδικασία, η αιτήσια ε, ε, των προϋπολογισμών δεν ελέγχεται ούτε από το Κοινοβούλιο ούτε από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Κανείς από όσους βρίσκονται εδώ δεν μπορεί να εξηγήσει το εκλογικό του σώμα πώς αυτή τη στιγμή υπολογίζεται το ύψος της, της εθνικής συνεισφοράς στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Ε, παλιά μας είχαν πει πως αυτά τα οποία προσπαθούμε να πετύχουμε είναι μια ουτοπία. Όσοι όμως στηρίζουν το status quo θα πρέπει ε, να να γνωρίζουν πως χρειάζεται μία μεταρρύθμιση, πως χρειάζεται μία μεγάλη αλλαγή έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μία γενικότερη συμφωνία και ξέρετε πως η συμφωνία μέσα στον επόμενο μήνα για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι ακρογωνίως λήθος για να πετύχουμε συμφωνία και στον προϋπολογισμό. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την περασμένη εβδομάδα είπε ο πρόεδρος Φαν Ρόμπα πως θα πρέπει να δούμε την ε, δημοσιονομική δυνατότητα που έχει η ζώνη του ευρώ. Και αυτό θα συζητηθεί στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Πρέπει να σας πω πως αυτό δεν μπορεί να σχετιστεί καθόλου με τις διαπραγματεύσει που γίνονται αυτή τη στιγμή για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πρέπει να σας πω το εξή. Για μα το θέμα αυτό παρεμβαίνει και παραμποδίζει την συζήτηση ε, μεν για τον προπολογισμό, αλλά παράλληλα συνδυάζεται απόλυτα μαζί της. Είπαμε πως θα πρέπει να έχουμε μια επιπλέον βοήθεια που θα προσφέρονται στα κράτη τα οποία κάνουν τη δύσκολη προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίνησης. Άρα λοιπόν τι κάνουμε. Επανασύσταση ε, του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση ή του Ταμείου Συνοχής για τα έσοδα. Επίσης, αν αυτό το νέο ταμείο προέρχεται από εθνική συνεισφορά, είναι προφανές πως ε, τα κράτη τα οποία χρηματοδοτούν το ταμείο αυτό θα βρουν κάποιο λόγο έτσι ώστε να παγώσουν ή να μειώσουν τη συνφορά τους ε, στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν λοιπόν θεωρείτε πως θα χρηματοδοτηθεί μέσω των ίδιων πόρων, τότε πρέπει να σας πω πως στην περίπτωση αυτή και πάλι θα πλήξετε τον ευρωπαϊκό Προπολογισμό και για το χρονοδιάγραμμα αντιμετωπίζουμε παρόμοια προβλήματα. Μα είπατε πω ε, είναι κάτι το οποίο θα αποφασίσουμε μελλοντικά. Ε, μην ανησυχείτε. Ναι, 1η Ιανουαρίου του 2013 δεν μπορώ να διαφωνήσω, Όμω αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε τεράστια κρίση χρέου και όπου συναντιέται συχνά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν μπορεί να συζητάει αποφάσεις που θα συζητηθούν μετά το 2020, δηλαδή μετά ε, τους ε, με τους επόμενους ε, προέδρους και με τους επόμενους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να ισχύσουν τα όσα είπα για τον προϋπολογισμό. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πως όλοι οι πόροι που μπορεί να δημιουργηθούν για να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη θα πρέπει να ενσωματωθούν στην τρέχουσα διαδικασία έγκρισης του κοινοτικού προϋπολογισμού. Και νομίζω ότι αυτή αποτελεί και τη βασική αρχή της ενότητας του προϋπολογισμού. Μπορούμε να έχουμε κάποια πίνακες ε, σε προσάρτημα, κάποιον επιπλέον ε, προπολογισμό σε παράρτημα για να χρηματοδοτήσουμε κάποιες επιπλέον δράσεις, αλλά θα πρέπει να, είναι, να μην γίνει ο προπολογισμό ένα ιστορικό μνημείο με το συμβολικό ποσό συνεισφοράς του 1% που δεν θα καλύψει τις επόμενες ε, ανάγκες μας ε, και να τις χρηματοδοτήσουμε με διακυβερνητικό τρόπο, ε, με τον τρόπο αυτό αποφεύγοντας κάθε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Ευχαριστούμε κύριε Λαμασούρ για το Συμβούλιο. Ο ε, Υπουργό Μαυρογιάννη, κύριο Μαυρογιάννη, έχει τον λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σα. Αξιότιμα μέλη, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι εισηγητές, ε, Αντιπρόεδρε κύριε Σεύκοβιτς, κύριε και κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να συμμετάσχω στην σημαντική αυτή συζήτηση. Ξέρουμε πόσο κρίσιμη είναι η συζήτηση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και θα πρέπει να δώσουμε την ε, απαραίτητη σημασία στην εμπρόθεσμη κατάληξη των διαπραγματεύσεων, μια και έτσι θα επιτραπεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, προχωρήσει στην εκτέλεση των δράσεων που ε, προβλέπονται. Εμείς συνεργαστήκαμε πολύ στενά με τα θέματα αυτά με το Κοινοβούλιο και πρέπει να σας πω πως είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στον Αλέν Λαμασούρ και στους δύο συνεισηγητές για τους φακέλους ε, στον κύριο Μπέγκε και στον κύριο Κάλφιν για την δέσμευση με την οποία προώθησαν αυτό το φάκελο και την αποφασιστικότητά τους έτσι ώστε να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να γίνει αποδεκτό και από τα δύο όργανα. Η Προεδρία της Κύπρου έχει αποδώσει ιδιαίτερη σημασία στο να συνεχίσουμε αυτή την τακτική της συχνής, των συχνών συναντήσεων μαζί σας και θα συνεχίσουμε μέχρι να βρεθεί κάποια συμφωνία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τον κύριο Ζαν Λουκ Ντεάν και την κυρία Άννη Γένσεν για τα όσα έχουν κάνει στο κομμάτι των εσόδων. Η Κυπριακή Προεδρία συνεργάζεται πολύ στενά με την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μια και το, ο φάκελος αυτός περνάει πια σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μέλη της έκαναν μεγάλα βήματα για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που δημιούργησε η χρηματοπιστωτική κρίση και αν ατενίσουμε το μέλλον πιστεύουμε ότι στο επόμενο πολιετές πρόγραμμα θα μας βοηθήσει για να ξεπερέσει με ε, διατηρήσιμο τρόπο η Ευρώπη την κρίση. Όλοι συμφωνούμε. Ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να έχει ένα καταλητικό ρόλο έτσι ώστε να δημιουργηθούν θέσεις εργασίες, να δημιουργηθεί ανάπτυξη σε όλη την Ευρώπη. Θέλουμε λοιπόν επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο και πιστεύουμε πως στο πολιετές αυτό πλαίσιο θα πρέπει να ε, μοχλευθούν οι ε, δαπάνες έτσι ώστε να στηρίξουν την ανταγωνιστικότητα, την σύγκληση ε, την απασχολησιμότητα και αυτά σε απόλυτη ευθυγράμμιση και συμμόρφωση με τους στόχους ε, του 2020. Όλοι γνωρίζουμε ποιοι είναι οι περιορισμοί που μας δεσμεύουν και σε μια περίοδο εξαιρετικής δημοσιονομικής πειθαρχίας είναι απαραίτητο το πλαίσιο αυτό να ε, αντικατοπτρίζει επίσης και τις προσπάθειες που καταβάλουν τα κράτη-μέλη να τυθασεύσουν τα χρέη τους και τα ελλείμματα στους προϋπολογισμούς έτσι ώστε αυτά να γίνουν βιώσιμα. Θα πρέπει να προσφέρει λοιπόν κάθε ευρώ προς θέμενη ευρωπαϊκή αξία και έτσι να προσπαθήσουμε η ποιότητα των δαπανών να βελτιωθεί στα πλαίσια αυτού του πολιτικού πλαισίου. Είδατε την αναθεωρημένη εκδοχή ε, του διαπραγματευτικού box που έχουμε ε, που παρουσιάσαμε στο Συμβούλιο το Σεπτέμβριο και στα πλαίσια του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων ε, στο Λουξεμβούργο την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε μια άτυπη συνάντηση όπου μιλήσαμε και με τους δικούς σας εκπροσώπους και όπου η η συνάντηση αυτή έδωσε πολλά αποτελέσματα. Το διαπραγματευτικό box θα παρουσιαστεί αναθεωρημένο την επόμενη εβδομάδα και εδώ θα δώσουμε μία σειρά αριθμητικών στοιχείων ε, έτσι ώστε να λύσουμε τα ποιοτικά θέματα που συνδέονται με κάποιους ε, τομείς δαπανών. Για τους ίδιους πόρους, να σας πω πως η Προεδρία χτες παρουσίασε ένα ανεπίσημο έγγραφο, ένα non-paper για να κινητοποιήσει τη συζήτηση κυρίως στα πολύ ε, ευαίσθητα θέματα των διορθώσεων. των καταλογισμών. Και επειδή γίνονται συζητήσεις αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σα δώσω ε, ένα πιο συγκεκριμένο στίγμα ε, για την πορεία που θα ακολουθήσουν οι συζητήσεις για το πολιτές πρόγραμμα, όμως εμείς η Κυπριακή Προεδρία εξακολουθούμε να πιστεύουμε πως από κοινού με το Κοινοβούλιο θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε με μεγαλύτερη βεβαιότητα ότι ποιοι θα είναι, ποιες θα είναι οι παράμετροι επί των οποίων θα βασιστεί μια συμφωνία. Ξέρετε πως έχει συγκληθεί στις 22 και 23 Νοεμβρίου μια έκτακτη ε, σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είπε πως ε, θα παραταθεί η συνάντηση αυτή όσο χρειαστεί. Η Κυπριακή Προεδρία στηρίζει τους στόχους αυτούς και με αυτά κατά νου εμείς συνεχίζουμε να καταβάλουμε ε, με κάθε ένταση τις προσπάθειες έτσι ώστε μέχρι την συνάντηση εκείνη του Νοεμβρίου να έχουμε κάποια μορφή συμφωνίας με εσά και με τα κράτη-μέλη. Παρακολουθούμε με πολύ προσοχή την ε, συζήτηση που γίνεται στα πλαίσια των εκθέσεων Μπέγκιο και Κάλφιν και θα μπούμε στη συζήτηση πιο συγκεκριμένα και αργότερα. Θέλω να τους ευχαριστήσω για τις εκθέσεις τους και να πω πως συμπεριλαμβάνουν πολύ σημαντικά θέματα τα οποία θα σχολιάσουμε και στα οποία θα επιστήσουμε την προσοχή των κρατών μελών για την ενδιάμεση λοιπόν έκθεση. Να ε, ευχαριστήσω λοιπόν και τον κύριο Λαμασούρ και την κυρία Γιέντσε να τους ευχαριστήσω για τον τρόπο με τον οποίο συνεργάστηκαν μαζί μας επίσης. Μέχρι σήμερα και ελπίζουμε πως θα συνεχιστεί αυτό το επίπεδο συνεργασίας ήταν πραγματικά εκπληκτικό και με τον κύριο Λαμασούρ και με όλη τη διαπραγματευτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δράτω με λοιπόν της ευκαιρίας για να σας ευχαριστήσω και προσωπικά κύριε Πρόεδρε, κύριε Σούλς για την προσωπική σας εμπλοκή και για την προσωπική σας συνδρομή. Για το γεγονός που είστε τόσο δεσμευμένος στο να πρικοδοτηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με το πιο σημαντικό μέσο το οποίο έχουμε στα χέρια μας για να ανταποκριθούμε και στις φιλοδοξίες μας που είναι η ανάπτυξη και η θέση εργασίας για την νεολαία έτσι ώστε όλοι να σεβαστούμε αυτό το συμβόλο τιμή μεταξύ γενναιών. Για να πετύχουμε τα καλύτερα λοιπόν αποτελέσματα για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο δεν αποτελεί μόνο προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας. Είναι μια κοινή προσπάθεια στην οποία εμπλέκονται και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο. Έτσι λοιπόν μετά την απονομή του Γραφείου Νόμπελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποδείξουμε στους Ευρωπαίους πολίτες πως μπορούμε να σταθούμε ενωμένοι ε, και να στηρίξουμε ένα ουσιαστικό τμήμα ε, του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να φανεί πως αποτελεί τμήμα της λύσης και να προσφέρει σε όλους τους πολίτες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα καλύτερο μέλλον. Ελπίζω να ακούσω και τις δικές σας απόψεις για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Μαυρογιάννη. Τώρα θα λάβει τον λόγο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Αντιπρόεδρος κ. Σεφτσοβιτς. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη. Πρώτα θέλω να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία να απαντήσω στην ε, ε, προσωρινή έκθεση του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου και να τοποθετηθώ. Συμφωνούμε ότι αυτή η πρόταση είναι η πιο σημαντική ως θέμα στο θεματολόγιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου διότι η απόφαση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα στείλει ένα σαφές μήνυμα προς τον έξω κόσμο ότι είμαστε σε θέση να επιτύχουμε με τη στρατηγική για το 2020 αν έχουμε επαρκή κονδύλια για να χρηματοδοτηθούν οι συναφείς πολιτικές και για να διαδραματίσουμε τον αναγκαίο ρόλο μας στη διεθνή σκηνή. Και έτσι βλέπουμε ότι για πρώτη φορά διαπραγματευόμαστε αυτά τα πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια υπό τη νέα συνθήκη. Και ο Γιάννου Λεβαντόφσκι και εγώ είμαστε υπέρμαχοι του να μπορέσουμε να δραθούμε τη ευκαιρία και να ασκήσουμε αυτά τα δικαιώματα και τι εξουσίε μα πλήρω. Θέλω να ευχαριστήσω την ε, Προεδρία για την δυνατότητα να υπάρξει καλή διαπραγμάτευση με το Ευρωκοινοβούλιο και την Επιτροπή και με την άτυπη ανταλλαγή απόψεων πριν από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων που ήταν πολύ θετική ευκαιρία. Εκεί διεξάγονται οι συζητήσει ε, για αυτά τα θέματα και από κοινού με τον Γιάννους Λεβαντόσκη. είμαστε υπέρ των προτάσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και υπέρ τη εμπλοκή ε, δραστήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μελετήσαμε την προσωρινή σα έκθεση σε λεπτομέρειε με ιδιαίτερη προσοχή και συμμεριζόμαστε την άποψη ότι είναι ένα προπολογισμό επενδυτικό επενδύσεων. Πρέπει να επαναλαμβάνουμε διαρκώ και αδιαλείπτω αυτό το μήνυμα διότι καμιά φορά το ξεχνάμε αυτό το μήνυμα μήνυμα στις διαπραγματεύσεις και στις ευρύτερες διαβουλεύσεις. Έχουμε σημαντικότατα επιχειρήματα στην πλευρά μας, διότι αναγνωρίζοντας το Συμβούλιο αυτό τον καταλητικό ρόλο για την δημιουργία θέσεων απασχόλησης ε, τον ε, Ιούνιο, αυτό το αποδεικνύει. Κάποιες παρατηρήσεις ε, Πρωτού δώσω τη σκητάλη στον συνάδελφο Γιάννου Λεβαντόφσκι που θα απαντήσει όλα τα δημοσιονομικά θέματα του προπολογισμού για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτον για τον όγκο του προπολογισμού. Επ' αυτού πιστεύω ότι είμαστε πεισμένοι ότι η πρότασή μας για το 1,08% του ΑΕΠ εκπροσωπεί ένα αξιόπιστο ποσοστό που θα βοηθήσει να σταθεροποιηθεί η χρηματοδότηση της κοινή ε, αγροτικής πολιτικής και της συνοχής και θα μας δώσει την ευκαιρία να έχουμε σημαντική αύξηση όσον αφορά τις προτεραιότητες ε, για τη στρατηγική του 2020. Εκτιμούμε ιδιαίτερα την εστίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για βελτιωμένη αναβαθμισμένη ποιότητα σε σχέση με τις δαπάνες. Διότι θέλουμε να πετύχουμε με αυτά τα κονδύλια ένα ποιοτικό άλμα και να πετύχουμε την ευρωπαϊκή πρόσθετη αξία. Θέλουμε να βελτιωθεί η αποδοτικότητα, η αποτελεσματικότητα και όσον αφορά τους μακροοικονομικούς όρους και προϋποθέσεις ε, Σημειώνω σε σχέση με τις παρατηρήσεις που έγιναν τα όσα ελέγχθησαν και θέλω να υπογραμμίσω ότι οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, συντάχθηκαν ως κίνητρο για τις διαθροτικές ε, μεταβολές και αλλαγές και να βελτιώσουμε με αυτόν τον τρόπο το δυναμικό μας. Δεν θέλουμε να υποστούν κυρώσεις τα κράτη-μέλη ή να διασφαλίσουμε καλύτερα ότι τα κονδύλια θα βοηθήσουν να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις και τα κενά τα οποία διαπιστώθηκαν. Τώρα, ιδιαίτερα όσον αφορά τις παρατηρήσεις έκθεση για τις διοικητικέ δαπάνε. Βεβαιώνουμε ότι το κατά 5% ε, μείωση των στελεχών είναι μια μεγάλη προσπάθεια που αναλαμβάνουμε και θα πρέπει να συνεισφέρει στην επίτευξη του τελικού στόχου. Και για το θέμα του συγχρονισμού Γνωρίζω ότι όλοι είμαστε πεισμένοι ότι πρέπει να ληφθεί μια απόφαση πριν από τα τέλη του 2012 ώστε να μπορέσουμε να αρχίσουμε με τις ε, αποτελεσματικές αυτές δαπάνες άμεσα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λεβαντόφσκι έχει τον λόγο. Επίτροπος παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, κύριε Υπουργέ, ξεκινώντας θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα των ιδίων πόρων. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί έδωσε μια νέα όθηση στις μεταρρυθμίσεις και στις συζητήσεις οι οποίες γίνονται με μια θα έλεγα διαφορετική μέθοδο αντίθετα με τον τρόπο με τον οποίο είχαμε ασχοληθεί στο παρελθόν με το θέμα. Να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Λαμασού ο οποίος διαπραγματεύτηκε το θέμα της, των αλλαγών στον τομέα των εσόδων και έδειξε τον δρόμο τον οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε για το μέλλον. Η ενδιάμεση έκθεσή σας περιλαμβάνει το βασικό μήνυμα της ενότητας του προϋπολογισμού. Η ενότητα αυτή μπορεί να ειδωθεί με πολλούς τρόπους. Αυτό το οποίο όμως έχει μεγάλη σημασία είναι να αντιληφθεί κανείς την ενότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Προϋπολογισμού, συγγνώμη, θα πρέπει οι δαπάνες και τα έσοδα να ενισχύουν ο ένας κλάδος τον άλλο και όχι να υπάρχουν τεχνητές αντιφάσεις ανάμεσά τους. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Είναι σημερινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να αδειοδοτήσει την ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα του φόρου για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ανάμεσα σε ορισμένα χώρη. Κάποιο σύστημα το οποίο αντικαθιστά ορισμένου στατιστικού τύπους ε, ε, φόρους ε, στον τομέα αυτό. Ακούμε από ορισμένε πρωτεύουσε όπως από το Λονδίνο ότι απαιτείται ένα σύστημα πιο δίκαιο και πιο διαφανές για τον τομέα ε, των ε, εσόδων και ακριβώς οι αιτήσει διορθώσεις αυτό επιτρέπουν και καθιστούν το σύστημα δίκαιο για όλους. Τώρα για τα οριζόντια θέματα, ξεκινώντας με το θέμα της ευελιξίας. Πράγματι υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, περισσότεροι περιορισμοί και γι' αυτό απαιτείται μεγαλύτερη ευελιξία. Ε, θα πρέπει όμως να δούμε τι είναι τα προβλεπόμενα και μη τα μη προβλεπόμενα συμβάντα. Πρέπει λοιπόν να αυξηθούν οι δυνατότητες στον τομέα της ευελιξίας και μέσω των ενδιαμέσων εκθέσεων. Υπάρχει επίσης και το θέμα του περιθωρίου για περιπτώσεις ανάγκης Μπορούμε σαν παράδειγμα με αυτόν τον τρόπο να καλύψουμε τις ανάγκες ε, του προγράμματος ε, οικονομικής ανάκαμψης. Αλλά βασιζόμεθα πάντα στο, ε, στα κεκτημένα που έχουν σωρευθεί κατά τη διάρκεια αυτής της δημοσιονομικής εντολής. Περιμένουμε περαιτέρω προτάσεις πάντως για να εκλεπτύνουμε ακόμα περισσότερο ε, τα θέματα αυτά μέχρι το 2020. Σχετικά με τα προγράμματα μεγάλης κλίμακας, μεγάλου μεγέθους, ο στόχος, τους είναι, στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε τη σωστή τους χρηματοδότηση. Πρέπει να συμφωνήσουμε λοιπόν στον τομέα αυτό. Συμφωνούμε επίσης και με το λεγόμενο στα γαλλικά «resta liquide», τα υπόλοιπα προς ρευστοποίηση. Πράγματι, στόχος της διαδικασίας είναι η ετήσια δημοσιονομική διαδικασία και η μόνη λύση για το θέμα αυτό του «resta liquide» είναι ε, πάντα το ετήσιο πλαίσιο του προϋπολογισμού και όχι τεχνητά μέσα τα οποία στην ουσία δημιουργούν προβλήματα και υπονομεύουν τις υποχρεώσεις. Και γενικά υπάρχει μια καθολική θα έλεγα εκπεφρασμένη βούληση για την απλούστευση του προϋπολογισμού των δημοσιονομικών διαδικασιών. Η κυρία Γκρέσλε ήταν μια πάρα πολύ σκληρή αλλά και ταυτόχρονα αποτελεσματική διαπραγματεύτρια και βοήθησε πάρα πολύ στο να πετύχουμε ε, τους στόχους που έχουμε ε, για την απλοποίηση των διαδικασιών. Φοβάμαι ότι υπάρχουν ε, ε, επιμέρους προγράμματα, πάρα πολλά, 57 προγράμματα, τα οποία αυξάνουν τις πιθανότητες γραφειοκρατίας. Το θέμα είναι λοιπόν εμείς να απλουστεύσουμε τις διαδικασίες και όχι βέβαια να τις καταστήσουμε πλέον αδύνατες. Έτσι μόνο θα μπορέσουμε να προσφέρουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϋπολογισμούς αξιοπρεπής από το 2014 μέχρι το 2020 αντίστοιχους με τις προκλήσεις. Ξεκινάμε τώρα με την συζήτηση σε σχέση με εισηγητές που έχουν ένα λεπτό από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές η σύστασή μου είναι να μην προσπαθήσετε σε αυτό το λεπτό να περιγράψετε το σύνολο του προπολογισμού. Δεν θα τα καταφέρετε και οι διαρμηνεί μα δεν θα μπορέσουν να σα παρακολουθήσουν. Ίσως να επικεντρωθείτε σε ένα σημαντικότερο σημείο για την κοινοβουλευτική σα επιτροπή. Αρχίζουμε με την κυρία Γιαννάκου, που είναι μια πεπειραμένη συνάδελφο και θα είναι σίγουρα σύντομη. Παρακαλώ, κυρία Γιαννάκου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο πολύ σωστά θα διατηρηθεί για μια επταετία. οι πληροφορίες όμως που φτάνουν σε εμά για τις διαπραγματεύσεις με το συμβούλιο δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικές. φαίνεται πως το συμβούλιο ζητά σημαντικές μειώσεις οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με την πραγματική κατάσταση της ένωσης καθώς και με την οικονομική κρίση διότι με έμεσο τρόπο το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο μπορεί να βοηθήσει. όσο αφορά στο κομμάτι global europe στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης η ευρωπαϊκή επιτροπή πρότεινε σωστά υψημένα κονδύλια και αυτά πρέπει να υπάρχουν διότι η ένωση πρέπει να παίξει το διεθνή της ρόλο και να ανταποκριθεί σε απρόβλεπτες πολιτικές ή άλλες καταστάσεις οι οποίες προκύπτουν καθημερινά. πρέπει να υπάρχει δηλαδή ένα εύρος και μια δυνατότητα να μπορεί η ένωση να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία και για τις διάφορες παρεμβάσεις που αφορούν στις δικαιούχους χώρες ιδιαίτερα σε αυτές που η δημοκρατία αποκαθίσταται αλλά και για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης αυτή καθ' αυτή. κύριε πρόεδρε το κοινοβούλιο οφείλει να στηρίξει συνολικά την αύξηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου όπως ακριβώς το κοινοβούλιο την έχει προτείνει και να επιμείνει γιατί το να παραμείνει στο πλαίσιο που θέλει το συμβούλιο θα αποτελεί και έναν απαράδεκτο συμβολισμό για τους πολίτες της ευρώπης για το πώ αντιλαμβάνεται το συμβούλιο της ευρωπαϊκής ένωσης την αντιμετώπιση των ουσιαστικών προβλημάτων αυτή. ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Γιαννάκου. Ο κύριος Γκέρεντ για την Επιτροπή ανάπτυξη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η μέθοδος του Μάλθους, σύμφωνα με την οποία δεν μπορούμε να ζούμε μέσα στην ευημερία ενώ άλλοι ζουν μέσα στη φτώχεια παρά μόνο τότε, είναι κάτι που έχει ξεπεραστεί πλέον. Η βοήθεια προς την ανάπτυξη γενικότερα είναι βασικό συστατικό του τρόπου λειτουργίας μας και γι' αυτό ακριβώς απευθύνουμε έκκληση στις κυβερνήσεις των κρατών μελών να, να εναντιωθούν σε αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι η βοήθεια για την ανάπτυξη είναι ένα εμπόδιο σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε. Αυτό δεν θα πρέπει να εμποδίσει τη δράση μας στα πλαίσια των ανθρωπιστικών παρεμβάσεων, ε, όπου βέβαια αποτελούμε τον πιο αποτελεσματικό θα έλεγα και τον σημαντικότερο πρωταγωνιστή στον κόσμο. Είμαστε σημείο βοήθειας και αναφοράς για αυτούς οι οποίοι δεν τα καταφέρνουν ακόμα στον υπόλοιπο κόσμο. Χθε στα πλαίσια της συζήτησης ε, για την Agenda for Change καθορίσαμε κάπως καλύτερα τις θέσεις μας και σήμερα θα πρέπει πρακτικά να πάρουμε αποφάσεις οι οποίες να μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες τα επόμενα χρόνια. Για την Επιτροπή Παγκοσμίου Διεθνούς Εμπορίου, ο κύριος Καμάρ, παρακαλώ. Thank you very much, Mr. Ευχαριστώ πολύ. Οι κυβερνήσει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να σφίξουν το ζωνάρι τους, να μειώσουν ελλείμματα, να μειώσουν χρέος. Αλλά η λύση εδώ μοιάζει να είναι να αυξήσουμε το χρέος και να ε, σπαταλήσουμε και άλλα λεφτά φορολογουμένων με σπάταλες ε, ενισχύσεις. Τώρα στην ε, ΙΝΤΑ εμείς ζητήσαμε να γίνεται μια καλύτερη χρήση των υπαρχόντων κονδυλίων έτσι ώστε οι μικροί ομιστές επιχειρήσεις Ευρώπης να έχουν τη δυνατότητα να εξαπλωθούν σε διεθνείς αγορές και να βοηθήσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες ε, να τα πάνε καλύτερα στη δική τους χώρα και να βελτιώσουν εκεί τη ζωή τους έτσι ώστε να μην εξαρτώνται τόσο πολύ από εμάς. Αλλά ξέρετε πως το πώς θα επιστρέψουμε στην ανάπτυξη είναι το πρόβλημα, όχι το πόσα θα δαπανίσουμε. Για να δούμε ε, πόσα από τα κράτη που βρίσκονται ε, στην ε, κορυφή των επιχειρήσεων που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Πού είναι η ευρωπαϊκή Google, πού είναι οι ευρωπαϊκοί ε, επενδυτέ και ερευνητέ που θα μα φέρουν στην κορφή αυτή. Ευχαριστώ κύριε Κάμαρα. Ο κύριο Μούλτερ για την Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού, παρακαλώ. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για την Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού, το πιο σημαντικό είναι τα κονδύλια αυτά να επενδυθούν, να χρησιμοποιηθούν με το σωστότερο τρόπο. Δηλαδή, με άλλα λόγια, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι αναμένουμε ότι το ελεγκτικό συνέδριο θα μπορέσει να δώσει μια θετική δήλωση αξιοπιστίας και όχι μια αρνητική δήλωση. Η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού θεωρεί ότι μια εθνική πιστοποίηση από τα κράτη-μέλη είναι απόλυτα αναγκαία τουλάχιστον από τα κράτη-μέλη πρέπει να υπάρχει η υπευθυνότητα για την δαπάνη, την διάθεση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα πιθανότατα θα έχουμε και την προαγωγή της ψήφισης ε, ώστε να μπορέσει να δημιουργηθεί αυτό το πλαίσιο δηλώσεων αξιοπιστίας από, από τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να ενθαρρυνθούν τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν με αυτή τη δήλωση αξιοπιστίας και πρέπει να υπάρξουν και κίνητρα που θα τους δίδονται προτιμησιακά κίνητρα εναντί άλλων χωρών. Ευχαριστώ. Για την Επιτροπή απασχόληση, η κυρία Μπερέ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το θεμέλιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση που τιμήθηκε από την Επιτροπή Νόμπελ είναι η αλληλεγγύη. Δεν υπάρχει αλληλεγγύη όμω χωρί χρήματα, δηλαδή χωρί προπολογισμό. Γνωρίζουμε ότι τα τελευταία 14 χρόνια οι προπολογισμοί εθνικοί αυξήθηκαν πιο γρήγορα από του κοινοτικού και τώρα το Συμβούλιο θέλει ε, ο, ο προϋπολογισμός της Ένωσης να μειωθεί πιο γρήγορα από τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Ταυτόχρονα ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ζητά εμείς να μην εγκαταλείψουμε το κοινωνικό μας πρότυπο. Άλλοι πιστεύουν ότι η πολιτική λιτότητα στην οποία πρεσβεύουμε είναι αντιπαραγωγική. Η πρώτη διαρθρωτική αλλαγή που πρέπει να γίνει λοιπόν είναι στον τομέα των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Δεν μου αρέσει αυτή η έκφραση αλλά σημαίνει κάτι. Ο βασικός μας πλούτος είναι η ποιότητα των ανδρών και των γυναικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει εμείς να προσπαθήσουμε να ορίσουμε με σωστό τρόπο τις δαπάνες στον τομέα των κοινωνικών και ε, θα πρέπει επίσης ε, τα χρήματα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας για τον κοινωνικό τομέα να τα χρησιμοποιήσουμε με σωστό τρόπο. Έτσι θα υπερασπιστούμε και το πρόγραμμα το οποίο θα βοηθήσει τους λιγότερο σε χαμηλότερη... Ευχαριστώ κυρία Μπερές για την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, η συνάδελφος κυρία Χέρτσογκ. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα αυτό το οποίο πρέπει είναι να αλλάξουμε την πολιτική μας και να είμαστε ενωμένοι. Πρέπει να δημιουργηθούν οι συνθήκες πλαίσιο για την ανάπτυξη. Πρέπει να δημιουργηθούν δομές που θα, θα μπορέσουν να προχωρήσουν την οικονομία μας. Χρειαζόμαστε και την ενιαία εσωτερική αγορά και σημαντικά βήματα. Με αυτά τα βήματα μπορούμε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως μέλος της Επιτροπής ΙΤΡΕ θέλω να τονίσω και να πω πόσο σημαντικό είναι αυτή την ανάπτυξη, σε αυτή την ανάπτυξη να επενδύσουμε. Χρειαζόμαστε πολιτικά μέτρα για την βιομηχανική ανάπτυξη. Δεν μπορούμε να δεχτούμε και να αφήσουμε πολιτικά προγράμματα όπως ε, ο Γαλιλαίος ε, να γίνουν θύματα του κανιβαλισμού άλλης χρήσης κονδυλίων. Χρειαζόμαστε τα προγράμματα αυτά. Χρειαζόμαστε και το πρόγραμμα για την Connecting Europe, ε, τη διασύνδεση της Ευρώπης. Χρειαζόμαστε θέσεις απασχόλησης για τους νέους επιχειρηματίες, για τους νέους γενικότερα είναι η μεγαλύτερη απώλεια αυτή της οικονομικής κρίσης, η απώλεια αυτής της νέας γενεάς. Πρέπει κάτι να κάνουμε οπωσδήποτε επιτέλους. Αγαπητοί Επίτροπε, θα σας υποστηρίξουμε στο εγχείρημά σας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Χέρσογκ. Για την ίδια Επιτροπή θα λάβει τον λόγο η κυρία Ματίας παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Στη συνεργασία με τους συναδέλφους, ιδιαίτερα όσον αφορά τον δημόσιο τομέα, ζητήσαμε ένα πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο που δεν θα ξεχνά την δημόσια υγεία και το περιβάλλον μέσα στην συγκυρία της κρίσης. Διότι αυτό γίνεται σε σχέση με τα κράτη-μέλη. Τα ξεχνάμε. Να υπάρξει χρηματοδότηση σε σχέση με τις προτάσεις ε, για την ε, ε, πολιτική αυτή στην Ευρώπη, για την κλιματική, κλιματολογική πολιτική. Ζητάμε κονδύλια πέρα από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την διασφάλιση και διατήρηση της φύσης και της βιοπικιλότητας στο πρόγραμμα LIFE. Ζητούμε επίσης την προστασία της, του τομέα των πολιτών πολιτική προστασία. Αυτά είναι σημαντικά για να ξέρουμε αν προχωράμε ή όχι μέσα στην κρίση. Και το ότι μιλάμε για την πολιτική, τους πολιτικούς προσανατολισμούς, αυτό που θέλουμε είναι να πάψει η λιτότητα, να υπάρξει αλληλεγγύη, να υπάρξει η κοινωνική αλληλεγγύη. Αυτό πρέπει να γίνει. Είναι εξαιρετικές οι περίοδοι που περνούμε, ξεχωριστές και πρέπει με ξεχωριστές πολιτικές ε, να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα πρέπει να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να κερδίσει η Ευρώπη σε αυτά τα στοιχήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ματίας. Τον λόγο τώρα θα λάβει για την Επιτροπή Μεταφορών ο συνάδελφος Σίμψον παρακαλώ. Σήμερα το πρωί εκφράζω ε, την Επιτροπή Τουρισμού και Μεταφορών και θα ήθελα να σεβαστώ ε, τις συμβουλές σας για δύο πολύ σημαντικά θέματα. Καταρχήν, πώς θα πρέπει να ενισχύσουμε ε, την απασχόληση και να βρούμε θέσεις εργασίας έτσι ώστε να ανακάμψει η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση σύμφωνα με τα όσα έχουμε στην ατζέντα του 2020 και επίσης πως οι υποδομές είναι απαραίτητες για να παραδώσουν σε αυτά τα πλαίσια αυτές τις νέες θέσεις εργασίας. Χαιρετίζουμε λοιπόν την πρόταση της Κομισιόν για το μηχανισμό Connecting Europe για τη διευκόλυνση αυτή που θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε αυτά που επιθυμούμε και έτσι ώστε να έχουμε υποδομές οι οποίες θα είναι βιώσιμες, διατηρήσιμες και επιτεύξιμες. Χρειαζόμαστε βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να δώσουμε μια ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία ε, στις μεταφορές και υποδομή στα κράτη-μέλη. Αλλά καμιά φορά υπάρχει μια έλλειψη συντονισμού ή επικοινωνίας μεταξύ Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών. Ως συμπέρασμα θα ήθελα να επαναλάβω πως η πρόταση της ε, ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής γίνεται δεκτή από τη δική μας Επιτροπή. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Κοβάτσεφ ε, για την Επιτροπή Περιφερειακή Ανάπτυξης. Αγαπητοί συνάδελφοι, αξιότιμοι επίτροποι, Στη δική μας Επιτροπή αποφασίσαμε πως η χρηματοδότηση για την πολιτική συνοχή θα πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον στα επίπεδα που είχαμε στην περίοδο 2007-2013 γιατί αυτό αποτελεί το ελάχιστο επίπεδο χρηματοδότησης ε, που θα καλύψει τις ανάγκες μας είναι το χαμηλότερο όριο κάτω από το οποίο δεν θα πρέπει να πέσουν οι κυβερνήσεις μας στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Θα πρέπει να επενδύσουμε σε μέσα τα οποία θα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη στην ανάπτυξη και στην ανάταξη των ε, περιφερειών της Ευρώπης και που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Μας είπαν πως χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Μη φανούμε υποκριτές. Εμείς ακούμε όλες αυτές τις εκκλήσεις για την περισσότερη Ευρώπη και παρόλα αυτά κάποια, ε, κάποια αρχηγοί κρατών ε, κυβερνήσεων αυτή τη στιγμή διαπραγματεύονται περικοπές σε αυτήν την περισσότερη Ευρώπη. Κάτι το οποίο θα υποσκάψει τους στόχους που έχουμε θέσει στα πλαίσια της στρατηγικής για το 2020. Σας απευθύνω εγώ μια έκκληση. Αξιότιμοι συνάδελφοι να στηρίξετε αυτή την απόφαση για το πολιετές πρόγραμμα του δημοσιονομικού πλαίσιο για το πίδι πει. Ε, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να μιλήσω εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Κοιτάξτε τι συμβαίνει σε ορισμένες χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ελλάδα ή ε, κοιτάξτε τι συμβαίνει σε φτωχές περιοχές ε, κάποιων πλουσίων χωρών όπως η Φιλανδία στην ανατολική της πλευρά. Τι θα κάνετε για αυτές τις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί σήμερα. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά την ερώτησή σας, λέει ο κ. Καρφίν, αλλά στον τομέα της ε, πολιτικής συνοχής θα ήθελα να πω ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τα διαθέσιμε τις διαθέσιμες πιστώσεις και οι δύο κατηγορίες χωρών μπορούν να βοηθηθούν από αυτά τα μέσα αλληλεγγύης χρήσιμα μέσα και για τις χώρες οι οποίες συνεισφέρουν περισσότερο στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να το εξηγήσουμε αυτό στους φορολογουμένους να πούμε ότι δεν υπάρχουν μόνο αυτοί που κερδίζουν και αυτοί που χάνουν, αλλά όλα τα εκατομμύρια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ωφελούνται από την πολιτική συνοχή. Ελπίζω να ήταν αυτή η ερώτησή σας. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Θα δώσω το λόγο για ένα λεπτό στον κύριο Δεκάστρο. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η Επιτροπή Γεωργίας ε, τις οποίας προεδρεύω και τις οποίες είμαι εισηγητής για την ενδιάμεση έκθεση, εξέφρασε την ε, πρόθεση, την, την απόφαση της ε, να μην παγώσει ο προϋπολογισμός σε ε, θεωρητικό επίπεδο, σε ονομαστικό επίπεδο, αλλά σε πραγματικό επίπεδο, με πραγματικούς αριθμούς και γι' αυτό υποστηρίζουμε την πρωτοβουλία Μπέγκε και Κάλφιν που έκαναν μια εξαιρετική προσπάθεια. Αυτό θα μας επιτρέψει να έχουμε μια ενωτική και ισχυρή θέση από πλευράς Κοινοβουλίου. Να υπογραμμίσω εν τω μεταξύ ότι ο, εφόσον υπάρξουν περικοπές στον προϋπολογισμό περαιτέρω, τότε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμφωνήσουμε για τις διαδικασίες μεταρρύθμισης όλοι οι συνάδελφοι από όλε τι πολιτικέ ομάδε δεν θέλουν να υπάρξει μια τελική ψήφο για τι μεταρρυθμίσει αν δεν διευκρινιστεί το θέμα του προπολογισμού. Ενό προπολογισμού που θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στι προκλήσει, τι οποίε επιβάλλει το μέλλον στη γεωργία τη Ευρώπη. Ο κύριος Φερέιρα, Επιτροπή Αλή. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η πρόταση δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 είναι μια μείωση σε σχετικούς όρους σε σχέση με το σημερινό πλαίσιο. Με αυτές τις προοπτικές δεν θα υπάρχει κοινωνική και οικονομική σύνοχη, αλλά μεγαλύτερη παρέκκληση. Και εδώ σε σχέση με τα, τις περικοπές του Συμβουλίου για θα πρέπει να υπάρξει αύξηση κονδυλίων για να είναι αποδεκτές οι προτάσεις. Χάσαμε σε σχέση με τις προτάσεις για τη θάλασσα 6 δισεκατομμύρια ευρώ και για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλλιείας και για τους πόρους της θάλασσας. Είναι ένα σημαντικότατο ποσό για κατά μέσο όρο αναέτος. Αυτή, αυτό το ποσό είναι ακόμα χαμηλότερο από εκείνο το οποίο είχε προβλεφθεί για το 2013, τελευταίο έτος του σημερινού, του, ε, σημερινού πλαισίου δημοσιονομικού πλαισίου. Πάντα χαμηλότερα αυτά τα ποσά από ό,τι είχαν προβλεφθεί. Δηλαδή, ακόμα και αν το σημερινό πλαίσιο είναι ανεπαρκέ, η πρόταση για το μελλοντικό δημοσιονομικό πλαίσιο είναι ακόμα χειρότερη. Όσον αφορά την ε, πρόταση αυτών των ισχνών κονδυλίων για, για άλλε χρήσει, αυτά όλα κάνουν αυτή την πρόταση ε, να μα δίνει επαρκή λόγου για την καταψηφίσουμε κάθετα. Ευχαριστώ. Λόκεγκατ, παρακαλώ, για την Επιτροπή Πολιτισμού. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε ως ε, εκπρόσωπος της ε, Επιτροπής Πολιτισμού είναι πραγματικά πολύ δύσκολο έργο σε μια περίοδο οικονομικής συγκυρίας λιτότητας και περικοπών να μπορέσουμε να πετύχουμε κάτι που θα λαμβάνει υπόψη τους νέους, τις ανάγκες τους και τον πολιτισμικό και πολιτιστικό τομέα. Ευτυχώς όμως επανειλημμένα και πάντα μπορούσαμε και μπορέσαμε να διαπιστώσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο αρμόδιος Επίτροπος πάντα υπέβαλε φιλόδοξες προτάσεις ε, και χαιρόμαστε γι' αυτό. Εδώ πρόκειται λοιπόν για την εκπαίδευση, κατάρτιση, για θέματα νεολαίας, ε, θέματα αθλητισμού, τομείς που πραγματικά σε αυτή την περίοδο περικοπών και λιτότητας ε, θα πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη και να προαθούν. Αυτό μας ικανοποιεί. Ωστόσο θέλω να απευθύνω έκκληση στα κράτη-μέλη που με θετικό τρόπο τοποθετήθηκαν στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όσον αφορά την υποστήριξη υποστήριξη που θα δοθεί. Αυτά όμως τα οποία θα αποφασίσουν και θα πούν οι Υπουργοί Οικονομικών θα πρέπει να αναμείνουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθούν αυτές οι διαπραγματεύσεις για να δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστώ. Ρότ Μπέρεν παρακαλώ στη συνέχεια. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, στο Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη έχω συχνά την εντύπωση, μου υπενθυμίζουν έναν παράν, εκείνο τη σάβρα της ε, Ινδονησίας ε, που έχει διχαλωτή γλώσσα. Είναι διχασμένες προσωπικότητες όμως. Θέλουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσουν όλο και περισσότερα έργα και περισσότερες εξουσίες. Το υποστηρίζουμε αυτό. Δεν θέλουν όμως να δώσουν τη δυνατότητα να έχει την ικανότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει επαρκή στελέχη για να επαρκέσει. Ακούγοντας τους συναδέφους από την Επιτροπή Γεωργίας, τον κύριο Ντεκάστρο, Επιτροπή Πολιτισμού, την έρευνα, την κοινωνική πολιτική, την περιφερειακή ανάπτυξη, τεράστια σημασία ΜΙΣΑ όλοι αυτοί για τις περιοχές μας και τις περιφέρειές μας και για τα κράτη-μέλη. Αυτό όμως που δεν κάνουν τα κράτη-μέλη είναι να λάβουν υπόψη ποιος θα πρέπει να εκπονήσει αυτές τις πολιτικές και να τις καλύψει. Ποιος θα εκπονήσει τροπολογίες και προτάσεις ώστε αυτά τα κονδύλια να υπαρκέσουν. Οι υπάλληλοι είναι και τα στελέχη που πρέπει να υπαρκούν και πρέπει να είναι αναβαθμισμένου επίπεδου αυτοί οι υπάλληλοι πολυπολιτισμικού ε, επίπεδου και πολιτισ... πολυσχηδούς χαρακτήρα ε, με τον περισσότερο θα έλεγα μεγαλύτερο πλούτο πολιτισμικό. Τι βλέπουμε όμως ότι κάνουν εδώ, περικοπές κονδυλίων. Αν δεν υπάρξει λοιπόν συνάδελφοι επαρκές δημοσιονομικό πλαίσιο δεν θα είμαστε σε θέση κανένα πολιτικό τομέα να καλύψουμε επαρκώς. Γι' αυτό ζητώ κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου να με ρημνήσετε η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, η πρόταση για, το, για τα στελέχη, για τους υπαλλήλου να γίνει δεκτή ώστε να έχουμε επαρκείς υπαλλήλου για τι ανάγκε μα Ευχαριστώ. Η απουσία της κυρίας Ολμάγερ, ο κύριος Τρασκόφσκι θα λάβει τον λόγο. Παρακαλώ. We have to keep the pressure up. Θα πρέπει να διατηρηθεί η πίεση μέσω των πολιτικών μας οικογενειών έτσι ώστε να σεβαστούμε τα χρονοδιαγράμματα και να συμφωνήσουμε αυτό το πι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση χωρίς τα μέσα που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη στην Ευρώπη και θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την αφετηρία. Δεν μπορούμε να υποσχεθούμε μεγαλύτερη Ευρώπη, περισσότερη Ευρώπη χωρίς τον αντίστοιχο προϋπολογισμό. Και τώρα βέβαια υπάρχει και το εξή παράδοξο. Θα πρέπει όλες αυτές τις φιλοδοξίες να τις εξυπηρετήσουμε με έναν ενιαίο προϋπολογισμό και θα πρέπει εμείς να επιφυλάξουμε την κατάλληλη δημοκρατική εξέταση όλων αυτών των δαπανών που θα πρέπει να ε, κρατηθούν μέσα στο σωστό δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν χρειάζεται εμεί να επανεφεύρουμε τον ε, τροχό. Θέλουμε να δώσουμε τη μάχη για ένα φιλόδοξο πολιτες δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά δεν μπορούμε να δώσουμε αυτή τη μάχη αν σκεφτόμαστε συνέχεια τι θα γίνει με άλλου προπολογισμού ή νέου θεσμού. Αυτό όχι μόνο θα αποδυναμώσουν τη δική μα πρόοδο, αλλά θα οδηγήσουν και σε ένα κατακαιρματισμό τη Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ζούμπερ έχει το λόγο από την Επιτροπή Ισότητας και Δικαιωμάτων των Γυναικών. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Στη συζήτηση σε σχέση με την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και την Ισότητα των Φύλων ομόφωνο ήταν το αποτέλεσμα. Η πρόταση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο δεν αντανακλά τη σπουδαιότητα της αύξησης των κονδυλίων που απαιτούνται και για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υποβαθμιστούν περισσότερο τα κοινωνικά δικαιώματα μέσα σε μια περίοδο κρίσης. Για την χρηματοδότηση των εξειδικευμένων πολιτικών για τα δικαιώματα των, των γυναικών αυτό που λέγεται και είναι ότι πρέπει να υπάρξει αναγκαία στήριξη και ενίσχυση των αναγκαίων προγραμμάτων όπως του προγράμματος Δάφνη. Επίσης ε, του προγράμματος ε, για τα δικαιώματα ηθαγένειας των δικαιωμάτων των πολιτών και να, υπάρξει, να υπάρξουν κονδύλια για την ισότητα των φύλων και για την διάσταση της ισότητας των φύλων. Για την εργασία αυτή που είναι κέρια σημασία και πρέπει να διασφαλιστεί. Για τα δικαιώματα των πολιτικών υπέρ των γυναικών συμβαίνει ό,τι και με τις άλλες πολιτικές. Μείωση των κονδυλίων και βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει εδώ πέρα σημαντικότατη μείωση όσον αφορά τους στόχους της κοινωνικής και οικονομικής ε, και περιφερειακής ε, συνοχής. Αυτός είναι ο τομέας που ήδη οδηγεί σε μεγαλύτερες παρεκκλήσεις, πράγμα που είναι ολέθριο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Έχετε μια ερώτηση αλλά για τον προηγούμενο μιλητή, οπότε προτείνω να προχωρήσουμε στον επόμενο. Οπότε μπορώ να δώσω ε, το λόγο στους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Καταρχήν ο κύριος Γκαρίγα εδώ για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω πως είναι άδικο να κατηγορείται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη συζήτηση αυτή απλώς ότι ζητάμε μια αύξηση ε, πόρων. Δεν θέλουμε αύξηση δαπανών, θέλουμε κάτι πολιτικό. Είναι μια συζήτηση πολιτική για τις οροφές των δαπανών και για τους πολιτικούς στόχους που εξυπηρετούν. Και το τμήμα των κοινών ε, πόρων ε, όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν για να χρηματοδοτήσουν τις πολιτικές προτεραιότητες τις οποίες ψηφίσαμε πολλές φορές ως στόχο ε, στην, ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και νομίζω πως αυτές θα πρέπει και να επικεντρωθούν στο πώς θα εξυπηρετήσουμε τους στόχους της Ατζέντα 2020 ανάπτυξη θέσης εργασίας. Είναι πολύ φυσιολογικό η συζήτηση να γίνεται γύρω από το πώς μπορούμε αυτές τις προτεραιότητες να τις δούμε στα πλαίσια των περιορισμένων πόρων που έχουμε λόγω χρηματοπιστωτικής κράσης κρίσης. Αυτό το οποίο ε, δεν έχει ε, καμία λογική είναι εμείς από μόνοι μας να μας βάλουμε μια τρικλοποδιά και να μην επιτρέψουμε η χρηματοδότηση που θα έχουμε να εξυπηρετήσει τους στόχους μας. Ξέρουμε πώς θα κάνει περικοπές στο Συμβούλιο, ξέρουμε πώς θα μειώσει την πρόταση ε, την οποία επέβαλε η Κομισιόν, η οποία έτσι κι αλλιώς είναι ανεπαρκής. Και αυτό λοιπόν θα πρέπει να επιμείνουμε προς τα δύο αυτά όργανα, πώς το ουσιαστικό είναι, εάν θέλουμε, εάν θα έχουμε ε, λιγότερα χρήματα στη διάθεσή μας, τότε χρειαζόμαστε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ευελιξία για τη χρήση αυτών. Γιατί ένας περιορισμένος προπολογισμό χωρίς ευελιξία θα μας δέσει τα χέρια. Η κυρία Τόγια για δύο λεπτά. Σοσιαλιστές. Ο προϋπολογισμός είναι θα έλεγα εμβληματικός για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μας δείχνει να καταλάβουμε τι θέλει να κάνει και τι κάνει σήμερα. Εμείς έχουμε να κάνουμε βασικές επιλογές ανάμεσα σε έναν προϋπολογισμό επιβίωσης, συρρήκνωσης, έστω και λίγο για όλους, ή σε έναν θαραλέο προϋπολογισμό στοχευμένων επενδύσεων για την απασχόληση, για τους νέους, για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ανάπτυξή της. Όλοι θα πρέπει να κατανοήσουν, όπως είπε και ο συνάδελφος Καλφίν ξεκάθαρα, ότι η Ευρώπη μπορεί να πετύχει σήμερα αυτά τα οποία δεν καταφέρνουν οι χώρες μέλη για την οικονομία, για την περιφερειακή ανάπτυξη, για την ανάπτυξη της υπαίθρου, για την επιχειρηματικότητα, για το καλό των πολιτών της οι μεγάλες ευρωπαϊκές επιλογές καταπνίγονται από κάποιες λογιστικές ε, λεπτομεριακές συζητήσεις στο εσωτερικό του Συμβουλίου και από την διαίρεση ανάμεσα στους καθαρούς εισφορείς και σε αυτούς οι οποίοι ωφελούνται λογιστικά. Αυτό είναι ψευδοπρόβλημα, είναι ψευδοδήλημα. Όλες οι χώρες ωφελούνται από την ανάπτυξη και από την οικονομική σύγκληση. Το Συμβούλιο προσπαθεί να δώσει αριθμούς σε αυτή τη φάση στα διάφορα τμήματα του προϋπολογισμού. Πόλεμος δηλώσεων, λήψεις ε, συγκεκριμένων θέσεων, δεσμευτικών από ορισμένε χώρες που δημιουργούν προβλήματα τελικά και δεν θα έλεγα κάνουν τίποτα άλλο από το να ενισχύουν το αντιευρωπαϊκό πνεύμα ορισμένων. Αυτή είναι μια λανθασμένη θέση που δεν βοηθάει την κατάσταση. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Ευρώπη είναι θα έλεγα σε ευάλωτη κατάσταση, η Ευρώπη σήμερα είναι ατελής και έχει ανάγκη από ανάπτυξη. Έχουμε σταθεροποιηθεί τόσο πολύ πια που είμαστε πλέον σε ύφεση. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε σωστές επιλογές για το πολιετές πλαίσιο. Ευχαριστώ κυρία Τόγια. Κυρία Γένσεν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Από πλευράς της ομάδας των φιλελευθέρων της Άλντε η έννοια της ελαστικότητας είναι μια πολύ σημαντική έννοια. Όμως πρόκειται επίσης και για νέους επιπρόσθετους ίδιους πόρους. Εχθές ήδη το ζήσαμε και σε αυτό το έγγραφο εμπεριέχεται επίσης ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες όσον αφορά το θέμα των ιδίων πόρων. Είναι ένα άδικο σύστημα, ένα σύστημα που πρέπει να αλλάξει οπωσδήποτε και προβλέπεται και αυτό. Ωστόσο ανησυχώ πρέπει να πω κάπως για το ότι από πλευράς της Κυπριακής Προεδρίας τηρούν κάτι άκαμπτα το οποίο θα έπρεπε να εγκαταλείψουν. Δηλαδή στον προϋπολογισμό θα πρέπει οι πραγματικές ανάγκες να αντανακλώνται, να αντικαθρεφτίζονται και όχι να σκεφτόμαστε τι πρέπει να έχουν ως εκροές τα κράτη-μέλη. Θέλουμε να υπάρξουν περικοπές, λέει, εξοικονομήσεις των κονδυλίων για την ε, έρευνα, για να προστατευτεί, λέει, το περιβάλλον. Και επανειλημμένα αυτό εκφράζεται με διάφορους τρόπους διότι οι Υπουργοί Οικονομικών θέλουν να έχουν επιστροφές ε, στο, στον κορβανά τους. Ωστόσο υπάρχουν έξι σημεία για τους ίδιους πόρους. Αυτό που θέλουμε είναι να επιτευχθεί ένα καλύτερο σύστημα το οποίο θα εισαχθεί και θα λειτουργήσει. Παρακαλώ αυτά τα έξι σημεία να ληφθούν υπόψη. Η κυρία Τρούπερ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε Λεβαντόφσκι, κύριε εκπρόσωπο του Συμβουλίου, πρώτα απ' όλα πρέπει να διαπιστώσω και να πω ότι συγκλονίζομαι με συγκλονίζει ο λόγος της ε, Κυπριακής Προεδρίας. Πόσο λίγο υπάρχει φλόγα στην Ευρώπη. Δεν το νιώθω ότι θέλετε να εργαστείτε υπέρ του μέλλοντος της Ευρώπης με τις προτάσεις σας μέσα σε αυτό το, την πρόταση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ζούμε στην Ευρώπη γνωρίζοντας ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να εξηγιάνουν τους προϋπολογισμούς τους. Από την άλλη πλευρά γνωρίζουμε ότι από κοινού ενωμένοι χρειαζόμαστε κίνητρα για την αηφορία στην ανάπτυξη. Πρέπει να καταπολεμήσουμε τις κλιματικές αλλογές αλλαγές, να προσαρμόσουμε την οικονομία και τις βιομηχανίες μας σε χαμηλές εκπομπές ρήπων, να δώσουμε κίνητρα και ελπίδα στους νέους. Αυτά δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε όταν συρρυκνώνουμε τον προϋπολογισμό και τα κονδύλια όπως γίνεται αυτό πολλαπλά. Είναι ένα λανθασμένο πολιτικό μήνυμα και δεν, είναι, δεν δίνει καθόλου ελπίδα για το ευρωπαϊκό μέλλον και πνεύμα. Και πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να ρυθμίζουμε τις οικονομικές αγορές και να διασφαλίσουμε όμως ταυτόχρονα την ε, ισότητα και την δικαιοσύνη. Δεν είναι δυνατόν πάντα μόνο οι φορολογούμενοι, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι να πληρώνουν για τα σπασμένα της κρίσης. Οι τραπεζίτες και οι τράπεζες, τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα και ε, ε, οι Ινστιτούτα πρέπει να πληρώσουν. Μόνο έτσι μπορούμε να διασφαλίσουμε την κοινωνική Ευρώπη και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτή την πολιτική που ακολουθήθηκε μέχρι σήμερα. Τώρα υποβάλλει προτάσεις ε, ο Επίτροπος ε, Λεβαντόφσκι να πληρώνουν λιγότερα τα κράτη-μέλη όταν θα ε, συμμετέχουν στο σύστημα χρηματοοικονομικών, τέλους χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Να καταλήξουμε σε μια win-win κατάσταση για τα κράτη-μέλη και το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον. Ελπίζω ότι θα κινητοποιηθεί και θα κινηθεί το Συμβούλιο προς αυτή την κατεύθυνση. Τελευταία παρατήρηση. Υπάρχει η ε, ε, ε, εντύπωση ότι υπάρχουν καλοί λόγοι για κίνητρα που θα δημιουργηθούν για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Όμως είναι αδιαχώρητος και αδιέρετος ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Δεν θα απεμπολίσουμε τα δικαιώματα δημοκρατικού ελέγχου του προϋπολογισμού και των δημοσιονομικών που είναι δικά μας δικαιώματα και εξουσίες μας. Σας διασφαλίζουμε ότι με εμπιστοσύνη θα υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας ώστε να υπάρξει μια δημοκρατική Ευρώπη όσον αφορά τα δημοσιονομικά και τον προϋπολογισμό. Ευχαριστώ. Ashworth, λεπτό παρακαλώ. Θα ήθελα να συγχαρώ και τους εισηγητές και να σας πω πως πολλά από τα όσα έχουν συμπεριλάβει στην έκθεσή τους εμείς μπορούμε να στηρίξουμε. Όμως υπάρχουν τρία σημεία στα οποία θα ήθελα να σταθώ. Καταρχήν στο μέγεθος του προπολογισμού. Είναι σημαντικό να δείξουμε και εμείς πώς κατανοούμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη. Άρα λοιπόν θα πρέπει να επιμείνουμε και εμείς στο πάγωμα στο 1%. Για τους ίδιους πόρους είμαστε ανοιχτοί σε διάφορες προτάσεις, αλλά δεν μας έχετε πείσει ούτε για τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ούτε για το θέμα του ΦΠΑ. Για την επιστροφή, να υπενθυμίσω σε όσους βρίσκονται εδώ ότι είναι μια μαθηματική εξίσωση το θέμα και δεν είναι συναισθηματικό ή πολιτικό ζήτημα. Ζήτημα. Οι προσπάθειες που έγιναν για την επίλυση της κρίσης ε, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών οικονομιών είναι αξιέπαινες, όμως επειδή είναι πολύ περιορισμένοι οι πόροι μας, θα έπρεπε ενδεχομένως να αξιολογήσουμε διαφορετικά τις προτεραιότητες χρηματοδότησης που έχουμε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Σίγουρα θα είναι δύσκολες οι αποφάσεις, αλλά οι επιλογές αυτές θα πρέπει να βασιστούν στο πώς μπορούμε να πετύχουμε πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Άσουαρθ. Επόμενος ομιλητής ο κύριος Κλούτε για δύο λεπτά. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, ένα θερμό ευχαριστώ προς τους δύο εισηγητές. Πιστεύω συνολικά η έκθεση αυτή είναι μια καλή τοποθέτηση γενικά του Ευρωκοινοβουλίου σε αυτή την έντονη αντιπαράθεση μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου και Συμβουλίου. Υπό το πρίσμα της κοινοβουλευτικής μου ομάδας θα ήθελα κυρίως να επιστήσω την προσοχή ότι η πολιτική περικοπών των τελευταίων ετών προφανώς απέτυχε. Αυτό συνδέεται με χώρες που ε, αντιμετώπισαν τέτοιες περικοπές, είχαν ε, κατάρρευση των ε, εσόδων, η φτώχεια αυξήθηκε όμως και βλέπουμε ότι το να συνεχιστεί αυτή η πολιτική στο μέλλον δεν είναι σωστό διότι βλέπουμε ότι ένα μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού επανεπιστρέφει στα κράτη-μέλη και σε σχέση με μέτρα λοιπόν υπέρ της ανάπτυξης και της έρευνας για αυτούς τους λόγους ε, δεν μπορούμε να δεχθούμε με κανένα τρόπο τέτοιου είδου περικοπέ. Ένα ιστορικό προηγούμενο και παράδειγμα θέλω να αναφέρω. Η χώρα από την οποία προέρχομαι, η Ομοσπονδιακή Γερμανία, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αντιμετώπιζε μια παρόμοια βαθιά κρίση. Είχαμε σημαντικότατη ε, υπερχρέωση κατά τις αρχές του, της του 50 και με το πρόγραμμα Marshall είχαμε σημαντικά κίνητρα και ενίσχυση με προγράμματα υποστήριξης ε, και αυτό βοήθησε να διαφύγει η Ομοσπονδιακή Γερμανία από αυτή την κρίση και να προχωρήσει στην οικονομική ανάπτυξη με το πρόγραμμα Marshall. Πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε λοιπόν να περικόψουμε και να συνεχίσουμε τις περικοπές. Πρέπει να μπορέσουμε να τονώσουμε με κονδύλια και να δώσουμε κίνητρα για να καταλήξουμε στην ανάπτυξη και να ε, ξεπεράσουμε την κρίση. Γνωρίζω ότι είναι περιορισμένος ο χρόνος μου. Θέλω να υποστηρίξω ρητά αυτά τα οποία ανέφερε η για και για το θέμα των ιδίων πόρων και για το θέμα των, του τέλους ε, του φόρου επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Υποστηρίζουμε αυτές τις προτάσεις ε, και θέλουμε και να πούμε ότι το τέλος χρηματοοικονομικών συναλλαγών είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Αν μπορέσουμε εμείς ως Κοινοβούλιο να το προαγάγουμε προς το συμφέρον μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτή η ενδιάμεση έκθεση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο περιέχει κάποια θα έλεγα θέματα πάρα πολύ σωστά όπως η ανάγκη να μείνουμε σε ένα στηρίξιμο και ευέλικτο επίπεδο των δαπανών και να χρησιμοποιήσουμε σωστά και με ευέλικτο τρόπο τους πόρους. Το θέμα είναι όμως πώς θα τα χρηματοδοτήσουμε όλα αυτά. Ο παρόν μηχανισμός δεν είναι βιώσιμος και δεν είναι δυνατόν να εισάγουμε νέες μορφές αντιστάθμισης και διόρθωσης για τα κράτη-μέλη. Η Ιταλία την τελευταία δεκαετία είχε ένα αρνητική επιστροφή για δέκα δις περίπου το χρόνο. Η Βόρεια Ιταλία πρέπει να στηρίξει μια χώρα η οποία πηγαίνει πραγματικά χάλια και μια Ευρώπη η οποία υπακούει αποκλειστικά στους Γερμανούς. Άλλες χώρες όπως η Γερμανία και η Ολλανδία έτυχαν θετικών διορθώσεων που θέλουν πάντα να διατηρήσουν. Δεν έχει νόημα αυτό. Τότε σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να κάνουμε και μια διόρθωση για τη Βόρεια Ιταλία, την περιοχή της Παντάνια. Και αυτό ε, δεν θα πρέπει να είναι εις βάρος βέβαια της υπόλοιπης Ευρώπης. Χαρτόγκ. Πρόεδρε, κύριε Λεβαντόσκη, εχθές είχαμε το θέμα του προϋπολισμού για το έτος 2013. Τώρα έχουμε το δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020. Απειλείται αρνησικυρία από πλευρά, βέτο από πλευρά τη Μεγάλη Βρετανία και από πλευρά των Ολλανδών παρόμοια. Θα πρέπει να καταστεί σαφέ ε, προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι τα εθνικά κοινοβούλια δεν μπορούν να απειλούνται από αυτήν, διότι τα εθνικά κοινοβούλια αποφασίζουν αυτοτελώ ε, για τα ευρωπαϊκά κονδύλια και όχι εσεί εδώ. Και θα πρέπει να πάψει πια να γίνεται λόγος για διαρκή δημιουργία υπηρεσιών οργανισμών που δεν, ε, ε, είναι, δεν εξυπηρετούν την υλοποίηση των στόχων και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει σε σχέση με αυτά τα κονδύλια όταν ε, αυτά θα ληφθούν υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βελτιωθεί η κατάσταση και με το δικαίωμα βέτο θα αλλάξει η κατάσταση. Ευχαριστώ κύριε Χαρτούγκ. Στη συνέχεια Μαρινέσκου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η έκθεση Burger Calfin αντανακλά και ε, υπογραμμίζει τις προτεραιότητες που εγκρίθηκαν από το Ευρωκοινοβούλιο μέσα στο πλαίσιο της έκθεσης Λαμασούρ. Είναι σημαντική, ε, ιδιαίτερη σημασία ο προπολογισμό σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης. Κάνουμε λόγο για ένα προπολογισμό για τις ε, την δημιουργία επενδύσεων σε σχέση με τα κράτη-μέλη και βλέπουμε ότι η ε, λιτότητα ε, που κυριάρχησε. Ωστόσο θα έπρεπε να υποστηρίζεται με καταλητικά μέτρα που θα είχαν αποτέλεσμα το να παγώσουμε το επίπεδο στις οροφές του 2013 δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να δεχθούμε. Και όταν ε, βλέπουμε το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αλλαγές μόνο αν θα υπάρξει μια γενική προσαρμογή και αναθεώρηση του γενικού συστήματος ιδιών πόρων και του ε, ΦΠΑ και του τέλους ε, χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Όσον αφορά τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η στρατηγική που ακολουθήθηκε από την ομάδα μας δίνει ε, μια πρόταση κάτω από τις οροφές του Κοινοβουλίου ως προοπτική και αν, όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο δεν μπορούμε να το δεχθούμε. Τώρα, για την καταψήφιση από τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου της πρόταση του Συμβουλίου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο αυτό θα είναι μεγάλη οπισθοδρόμηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η είναι απόφαση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Όλοι οι Ευρωβουλευτές θα πρέπει να συμμετάσχουν και να εμπλακούν ώστε έτσι να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις για πολιτικά θέματα οριζόντιου, εγκάρσιου χαρακτήρα στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει προσθέτες αλλαγές να γίνουν όσον αφορά τα κράτη-μέλη. Η κυρία Χάουγκ, ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. <clears throat> Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, κάνοντας λόγο για το επόμενο δημοσιονομικό ε, πλαίσιο και για τις ε, πολιτικές μας ε, όταν συζητούμε για αυτά και υπάρχει αντιπαράθεση, αυτό είναι η μία όψη του, μετα, του νομίσματος, οι δαπάνες. Από την άλλη πλευρά πρέπει να αναδιαμορφωθεί η άλλη όψη του νομίσματος, τα έσοδα. Εδώ και 20 χρόνια ζητεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα πιο διαφανές, πιο δίκαιο και πιο αποτελεσματικό σύστημα ιδίων πόρων. Τώρα για πρώτη φορά μπορούμε να δώσουμε ιδιαίτερη πίεση ε, σε, αυτό το, ε, σε αυτή την απέτησή μας. Ζητήθηκε από πλευρά της Επιτροπής ε, ΣΟΥΡ η κατάργηση όλων των επιστροφών και η δημιουργία ενός ενιαίου ολοκληρωμένου προϋπολογισμού απόλυτα ανεξάρτητου από εισφορές κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόνο εν μέρη έλαβε υπόψη αυτές τις προτάσεις. Πρότεινε μια αλλαγή του συστήματος ΦΠΑ εμείς υποστηρίζουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακόμα και αν είναι μια σε κατά 40% μεταρρύθμιση μόνο. Είναι όμως ένα βήμα έστω, ένα βήμα προς την ορθή κατεύθυνση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε το βραβείο Νόμπελ ε, Ειρήνης ε, ως ε, ανταμοιβή Μπορεί όμως να υπάρξει πρόοδος μόνο όταν υπάρξει αναθεώρηση του συστήματος ιδίων πόρων και όταν πάψει πια να ισχύει το σύστημα καθαρών εισφορέων και καθαρών αποδεκτών. Όταν συμβεί αυτό τότε θα μπορέσουμε να έχουμε ένα σαφές πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρόσθετης αξίας και η, μικρόνια στην αντιπαράθεση θα πάψει πλέον να υπάρχει. Ο κύριος Λάιον για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Επίτροπε. Οι συνάδελφοί μου, φιλελεύθεροι δημοκράτες από το Ηνωμένο Βασίλειο και εγώ υποστηρίζουμε τις προτάσεις που γίνονται εδώ σήμερα. Πράγματι ήδη οι πόροι θα πρέπει να επιτρέψουν στην Ευρώπη να αυξήσει τους πόρους της και να μειώσουν τις εθνικές συνεισφορές. Είναι ένας έξυπνος τρόπος έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τις δαπάνες και να καλύψουμε τις ανάγκες για τον επόμενο χρόνο παρά να επιστρέφουμε προς τα κράτη-μέλη τις συνεισφορές τους. Έτσι θα στηρίξουμε και τη στρατηγική 2020 και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ανάπτυξη. Το 2017 θέλουμε πραγματικά έναν σωστό προϋπολογισμό, ισολογισμένο και έτσι θα μπορέσουμε ε, να καταπολεμήσουμε την λιτότητα και να προωθήσουμε την ανάπτυξη. Στη δική μου χώρα ε, τα χρήματα για την κοινωνική κάλυψη έχουν μειωθεί και δεν υπάρχουν δυνατότητες ανάπτυξης και δεν υπάρχει φυσικά δυνατότητα στήριξης επιπλέον του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Εγώ θα ήθελα ένα προϋπολογισμό να αντικατοπτρίζει τις σκληρές ε, στιγμές που ζουν οι ε, κυβερνήσεις των κρατών μελών. Ένας μικρότερος προϋπολογισμός αλλά πιο ευέλικτος για να καλύψουμε τις βασικές μας προτεραιότητες. Ευχαριστώ κύριε Λάιον Τσουμάνσκι. Ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ότι τα επιχειρήματα σε αυτή τη συζήτηση είναι πολύ καλά γνωστά έχουμε υπέρμαχους ενός ε, ε, μικρότερου προϋπολογισμού που λένε ότι πρέπει να υπάρξουν περικοπές. Άλλοι που είναι υπέρ μεγαλύτερου όγκου χρηματοοικονομικού και κονδυλίων λένε ότι μόνο έτσι με μεγαλύτερες δαπάνες μπορούμε να έχουμε μόχλευση που θα είναι αποτελεσματική. Εμένα με ενδιαφέρει κάτι τελείως διαφορετικό. Πώς είναι δυνατόν οι συντηρητικοί και οι σοσιαλιστές σε αυτή, σε αυτή την Ευρωβουλή να κάνουν λόγο για ένα ευρύτερο προϋπολογισμό. Όταν τα κόμματα στην ε, Αυστρία, Σουηδία, Γερμανία Γερμανία, ακόμα και Γαλλία επιθυμούν και ζητούν την μείωση των κονδυλίων του προϋπολογισμού. Δεν είναι πολύ εύκολο για τους σοσιαλιστές και τους συντηρητικούς να απαιτούν μεγαλύτερα κονδύλια και μεγαλύτερο προϋπολογισμό όταν γνωρίζουν ότι το Συμβούλιο τα πολιτικά αυτά συμφέροντά τους τα διασφαλίζει με περικοπές από την άλλη πλευρά. Ε, λοιπόν τότε το Ευρωκοινοβούλιο μπορεί πραγματικά να υποστεί μεγάλη ζημιά στην αξιοπιστία του και πραγματικά να γελιοποιηθεί με μια τέτοια πολιτική και να απολεστεί η αλληλεγγύη με ένα τέτοιου είδους θίασο και θέατρο. Σας ευχαριστώ η κυρία Σεν. Τονίζει ότι τα δισεκατομμύρια τα οποία δαπανώνται έχουν ε, κάποια αποτελέσματα. Το 2007 η ανεργία ήταν 7,3%. Σήμερα είναι 10,5% εκεί έχει φτάσει. Στην Ισπανία ε, μία από τους μεγαλύτερους αποδέκτες ε, χώρα η άνεργη είναι 25% ως ποσοστό. Το ΑΕΠ ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέμεινε πολύ ε, σε συμπιεσμένα επίπεδα. Να μην ξεχνάμε ότι το ελεγκτικό συνέδριο δεν εξέδωσε για τις δαπάνες ε, μια συνολική εγγύηση, μια ε, δήλωση αξιοπιστίας. Έχουμε γενικά μια αποτυχημένη πολιτική και βλέπουμε σε σχέση με την στρατηγική του 2020 τα προβλήματα. Η απασχόληση προέρχεται από νέες θέσεις απασχόλησης στη βιομηχανία τη μείωση της ε, γραφειοκρατικής επιβάρυνσης. Ε, πρέπει να υπάρξει ε, από πλευράς των πολιτικών μια, ένα είδος κούρεμα ώστε να μην υπάρχουν περιττές δαπάνες. Στη συνέχεια, Βάντερ Στούπ παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εμείς εδώ θέλω να πω ότι ζητούμε περισσότερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα 500 ε, εκατομμύρια ευρώ για την Ολλανδία δεν καταφέρνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τηρήσει τα υπεσχημένα δεν πρέπει να ξεπεράσει ε, λέει τα όρια και αυτό είναι ένα σφάλμα ένα σφάλμα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ολλανδία σχηματίζεται μια νέα κυβέρνηση. Πρέπει να ε, οδηγηθεί σε περικοπές, θα υπάρξουν περικοπές και βλέπουμε ότι σε σχέση με τα κονδύλια που απαιτούνται από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουμε 500 εκατομμύρια περισσότερα. Δεν τηρούνται λοιπόν τα υπεσχημένα. Είναι μια διχασμένη στάση, διχαστική στάση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά τούτο λοιπόν ζητώ να υπάρξει δικαίωμα από τα κράτη-μέλη. Στη συνέχεια η κυρία Χούμπνερ. Για του κινδύνους στους οποίου αναφέρθηκα στις διαπραγματεύσει καταρχήν η απόφαση για το ΠΔΠ. Αν δεν αποφασίσουμε τον Νοέμβριο, πώς θα εξηγήσουμε στου ε, πολίτες πως δεν θα αποτελέσει προπολογισμό Ευρωπαϊκή Ένωση, τον καταλήτη για τη δημιουργία θέσεων εργασία. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να μπορούν να δηλώσουν πως απερίφραστα πως προϋπολογισμός θα υπάρχει παρόλο που μπορεί να έχουμε κάποιες ε, περιπτώσεις άρνησης έγκρισης γιατί η νομική βάση το επιτρέπει για τις ε, διαπραγματεύσεις, ναι, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται. Μιλάμε για τις ε, δαπάνες, θα πρέπει οι διορθώσεις να είναι διάφανες και ελάχιστες. Σήμερα ξεκινάει η συζήτηση και θα ήταν ανεύθυνο να προχωρήσουμε σε εθνικές διορθώσεις που θα είναι όλο και πιο πολλές. Σίγουρα το υπάρχον σύστημα ΦΠΑ ε, δεν είναι εύκολο να αντικατασταθεί ίσως τελικά καταλήξουμε σε γνήσιους ίδιους πόρους που θα οδηγήσουν σε, μια μεταρρυθμιστική, σε ένα μεταρρυθμιστικό καταιγισμό στο μέλλον. Κάτι το οποίο θα μπορούσε να αποβεί επικίνδυνο για την ε, πολιτική συνοχής δεν θα πρέπει να αποκλίνουμε από το βασικό στόχο που είναι η επένδυση στην ανάπτυξη αλλά και μείωση των εθνικών και περιφερειακών αποκλήσεων. Θα πρέπει λοιπόν την μεθοδολογία του Βερολίνου να τη σεβαστούμε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Χούμπνερ. Θα περάσουμε τώρα λοιπόν στην επόμενη διαδικασία στο Catch the Eye. Ο κύριος Νικολέσκου πρώτος. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να συμμετάσχω στη σημερινή συζήτηση γιατί έχουμε την τροπολογία 72 την οποία στηρίζουν πολλοί συναδελφοί για τις άμεσες ενισχύσεις στη Γεωργία γιατί πιστεύουμε πως εδώ θα πρέπει να υπάρξει σύγκληση ε, με τον τρόπο με τον οποίο καταβάλλονται αυτές οι άμεσες ενισχύσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί έχουμε τα δύο συστήματα ε, τα οποία ε, νομίζω δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα και θα θέλαμε για τις ενιαίες ενισχύσεις το σύστημα να ισχύει με δίκιο και παρόμοιο τρόπο για όλους. Νομίζω ότι στο ψήφισμα σήμερα, στην απόφαση σήμερα, το Κοινοβούλιο δίνει μια πραγματική εντολή για να συνεχίσουν διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο και καλό θα ήταν η εντολή αυτή να συμπληρωθεί με τις προσδοκίες που έχουμε για περισσότερη ανάπτυξη στην Ανατολική Ευρώπη. Κύριε Σταπάς είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ. Η συνάδελφος κυρία Γιούτα Χάουγκ σωστά και δίκαια ανέφερε αυτό αυτή την υπόθεση. Αν ήταν εδώ η Επιτροπή του, ε, που απονέμει το βραβείο Νόμπερ, ποτέ δεν θα το είχαμε πάρει οι χώρες ε, καθαροί εισφορείς και οι χώρες αποδέκτες διαφοροποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν εντάσεις μεταξύ των χωρών εισφορέων και χωρών αποδεκτών. Αναφέρθηκε από πλευρά ε, του Επιτρόπου ότι αυτός ο προϋπολογισμός θα μπορούσε και θα έπρεπε να είναι ένας προϋπολογισμός εσόδων και προ, ε, προϋπολογισμός εξόδων δαπανών. Αν δει κανεί όμως τις μελλοντικέ προοπτικές είναι ζωφερές, ιδιαίτερα όσον αφορά τις εσωτερικές δομές. Για τα νέα κράτη-μέλη είναι η μεγαλύτερη πρόκληση αυτή, διότι από το Ταμείο Συνοχής και από τα διαρθωτικά ταμεία παίρναμε πολλά κονδύλια και μπορούσαν έτσι να διασφαλιστούν οι επενδύσεις που ήταν αναγκαίε. Θέλω να επιστήσω την προσοχή στην Ουγγαρία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ, με πολύ αρνητικό τρόπο σχεδίασε τα πράγματα. Δεν ε, ολοκληρώθηκαν μελέτε και μπορεί να απολέσουμε 30% των κονδυλίων συνοχή. Ευχαριστώ. Βλάσακ, ευχαριστώ ένα από τα σημαντικότερα σημεία, σημεία για τη διαπραγμάτευση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου είναι η συμφωνία για την κατανομή των κονδυλίων. Η Βερολίνιος μέθοδος που χρησιμοποιείται από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 για την κατανομή αυτών των κονδυλίων είναι μια πολύ καλή συμβιβαστική λύση. Με μεγάλη ανησυχία βλέπω τώρα να υπάρχουν συζητήσεις για την μείωση των συντελεστών για κράτη-μέλη που έχουν περάσει πάνω από το ε, μέσο όρο του ε, ΑΕΠ που απαιτείται. Θα ήθελα να απευθύνω έκκληση στην Κυπριακή Προεδρία να μην γίνουν τέτοιες αλλαγές, τέτοιες μεταβολές που θα οδηγούσαν στη μείωση των κονδυλίων για λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Υποστηρίζοντας την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη σημαίνει να επικεντρώνουμε τους περιορισμένους πόρους μας στις περιοχές και περιφέρειες που τους χρειάζονται περισσότερο. Ο κύριος Κέλλη παρακαλώ. Νομίζω ότι η συζήτηση πρωινή σήμερα στην ουσία μπορεί να οριστεί σαν μια έκκληση και μια πρόκληση για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πρώτον να ρυθμίσει τα δημοσιονομικά μέχρι το τέλος του χρόνου και δεύτερον αυτό που είπε ο κύριος Μπόγκ. Αν θέλουν πράγματι να υπάρξουν μειώσεις θα πρέπει να τις τεκμηριώσουν ε, γιατί υπάρχουν πολλά που πρέπει να καλυφθούν όπως η κοινή αγροτική πολιτική, η πολιτική συνοχή, η Ατζέντα 2020 και όλα τεκμηριώνονται μέσω της προσθήκης ε, αξίας. Αν δεν υπάρχει προστιθέμενη αξία είναι πάρα πολύ δύσκολο να δεχτούμε τα επιχειρήματα αυτά. Δεύτερον, να πω ότι το δεύτερο κομμάτι των συζητήσεων σήμερα για τους ιδίους πόρους θέλω να συγχαρώ τις χώρες που, έχουν χρησιμοποιήσει ε, την, που θα χρησιμοποιήσουν μέσω ενισχυμένης συνεργασίας ε, τον φόρο για τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Εφόσον χρησιμοποιηθεί σωστά ο φόρος αυτός είναι κάτι που θα βοηθήσει πάρα πολύ στην ε, μείωση της πίεσης στο μέλλον. Κύριε Σάλβες. Ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς μπορεί να διασφαλίζει το Συμβούλιο ότι μπορεί η συνέχεια να διασφαλιστεί με δίκαιο τρόπο όταν στη συνέχεια λέει ότι αναγνωρίζει η Προεδρία ότι είναι αναπόφευκτο το τελικό επίπεδο των δαπανών να πρέπει να μειωθεί και ότι αυτές οι κατηγορίες θα πρέπει να υποβληθούν σε μια προσπάθεια μείωσης ξε, ξεχνάνε την ε, ε, στρατηγική της Λισαβόνας να είμαστε η πιο δυναμική οικονομία παγκόσμια μέχρι ε, την, τους, τα τελικά όρια που θέσαμε ξεχνάνε τη στρατηγική για το 2020 είναι μόνο λόγια και να περιεχομένου και το ποσοστό της ανεργίας που έχει αυξηθεί και σε σχέση με την, το ΑΕΠ για την ανάπτυξη και την έρευνα και όταν βλέπουμε ότι έχουμε μείωση των κονδυλίων και βλέπουμε αύξηση των, ε, του αριθμού των ατόμων που ζουν κάτω από τη φτώχεια. Δεν είναι λοιπόν μόνο ένας προϋπολογισμός δαπανών. Είναι ένας προϋπολογισμός ε, για τις επενδύσεις και στην έρευνα που είναι απόλυτα αναγκαίες ε, από πλευράς των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Ο κύριος Πάσκα παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Πού βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακρογωνιαίος λήθος είναι η αξία που προσφέρουν και η χρηματοδότηση μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολλούς ε, θεσμούς. Είναι μόνο μέσω των Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων που οι λαοί της Ευρώπης μπορούν να αποφασίσουν πώς, ε, ποιο κομμάτι ε, των πόρων τους θα διατηθούν μέσω του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Και αυτή τη στιγμή πιέζουμε όλους να κάνουν εξοικονομήσεις. Άρα λοιπόν και εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ξαναξιολογήσουμε τις προτεραιότητες μας και να τις τροποποιήσουμε ανάλογα για να αντιμετωπίσουμε και την οικονομική πραγματικότητα. Θα πρέπει να ψάξουμε μοντέλα τα οποία θα προχωρήσουν σε μια ανακατανομή πόρων στα πλαίσια του τρέχοντος προϋπολογισμού και θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε ε, έργα τα οποία ε, επιτρέπουν την ανάπτυξη και όχι αυτά τα οποία δεν θα ε, στηρίξουν την ανάκαμψη. Ο κύριος Σικύρης και ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Το προτινόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι ισχνό πραγματικά και ανεπαρκές σε μια περίοδο ε, συγκυρίας οικονομικής όπου πρέπει να υπάρξουν περικοπές ε, δεν είναι δυνατόν να δικαιολογηθούν επιπρόσθετες περικοπές ε, και όταν βλέπουμε ότι δεν ανταποκρινόμαστε στους στόχους που για να καλυφθούν εδώ δεν πρέπει να υπάρξουν περικοπές αλλά αυξήσεις. Είναι η λάθος έκθεση και σε σχέση με τις εκτιμήσεις αυτές πρέπει να πούμε ότι ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται σύμφωνα με παλαιές ανεδαφικές βάσεις υπολογισμού που δεν είναι πλέον επίκαιρες. Ο δεύτερος πυλώνας για παράδειγμα βλέπουμε ότι ο βασιζόταν σε σχέση με κάποια κριτήρια για τη συνοχή. Ο δεύτερος πυλώνας ε, ωφελούσε ιδιαίτερα τις ε, ε, περιφέρειες, τις γεωργικές περιφέρειες, λιγότερο όμως τους γεωργούς. Αν υπήρχε λοιπόν μια τέτοια σύνδεση θα έπρεπε αυτή να ληφθεί υπόψη. Παρακαλώ, επόμενος ομιλητής. <laughs> Η κυρία Κλέμπερ, σας ευχαριστώ. Έχουμε μπροστά μας ένα έγγραφο το οποίο είναι πολύ χρήσιμο σε σχέση με την υλοποίηση των σημαντικότερων στόχων ε, στο μέλλον. Θέλω να δραχθώ αυτή τη ευκαιρία για να αποστείλω ένα μήνυμα απόλυτα σαφέ προ το Συμβούλιο και προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε αυτή την περίοδο κρίση, τα κονδύλια του προπολογισμού πρέπει να υπαρκούν ώστε να διασφαλίζεται η ανάπτυξη και η συνοχή. Και γι' αυτό πρέπει να είναι ένα μέσο, ένα εργαλείο για το συντονισμό τη επίτευξη των στόχων που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διασφάλιση των ε, προγραμμάτων και των επενδύσεων για την ανάπτυξη, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων που σε αυτή την περίοδο υλοποιούν τα διάφορα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ τον κύριο Φλάσακ και τους άλλους συναδέρφους ε, που τοποθετήθηκαν επειδή υπογράμμισαν τις ανάγκες των περιοχών, των περιφερειών, των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών όπως για παράδειγμα στη Σλοβενία που μπορούν να ε, ζημιωθούν με αυτή τη μείωση. Ο κ. Παπα-Νικολάου παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε όλοι συμφωνούμε σήμερα ότι το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο αποκτά κεφαλαιώδη σημασία για την επόμενη περίοδο μια περίοδο που την χαρακτηρίζει όπως σήμερα όλοι ανέφεραν ε, υψηλά νούμερα ε, ανεργίας ε, ύφεση αρνητική ρυθμή στην ανάπτυξη. και ενώ λοιπόν όλοι αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες που έχουμε προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονό ότι για την κατανομή των κονδυλίων και αναφέρομαι ιδιαιτέρω στο ταμείο συνοχή και στο ταμείο περιφερειακή ανάπτυξη και θα ήθελα μια απάντηση γι' αυτό από την επιτροπή και από την προεδρία αν είναι δυνατόν ότι λαμβάνουμε υπόψη μα τα οικονομικά μεγέθη και το κατακεφαλήν εισόδημα στι περιφέρειε ε, από τα έτη. 2009 2009-2010. διευκρινίζω ότι αυτό οδηγεί σε μεγάλε αδικίε από τότε μέχρι σήμερα είχαμε πολύ ραγδαίε αλλαγές και δυσμενείς εξελίξεις στην ελλάδα για παράδειγμα η οικονομική συρρήκνωση έφτασε περίπου στο 18,4 ένα νούμερο δηλαδή αντίστοιχο με αυτό που είχε η γερμανία και η αμερική στην περίοδο της μεγάλης ύφεση. αντιλαμβάνεται η επιτροπή αυτή την αδικία; ξέρω ότι έχει τεθεί αυτό και από την ελληνική κυβέρνηση. θα έχουμε κάποια εξέλιξη στο θέμα αυτό; ευχαριστώ πολύ. Κυρία Thank um, Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλο και περισσότερο πρέπει να είναι το Κοινοβούλιο της Ευρώπης, όχι μια συλλογή κοινοβουλίων των κρατών μελών. Και συγχαίρω τους συναδέλφους Καλφίν και Μπέργκερ γιατί με την έκθεσή τους αντικατοπτρίζουν την πραγματική ευρωπαϊκή διάσταση. Μέχρι τώρα συζητούσαμε για τη διάσταση ανάμεσα σε αυτούς που πληρώνουν και σε αυτούς οι οποίοι λαμβάνουν. Θα πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε τις δυσκολίες των κρατών μελών. Αλλά θα πρέπει επίσης να πούμε ότι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι προϋπολογισμός ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Οι εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών επιτροπών το είπαν αυτό. Να πω προς τους συναδέλφους ότι τα χρήματα αυτά τα χρειαζόμαστε και για την κοινή αγροτική πολιτική. Ακούμε βέβαια το τι λένε τα κράτη-μέλη, ε, κάποια από αυτά που θεωρούν ότι αντιμετωπίζονται με κακό τρόπο λόγω των διαφορών στο σύστημα πληρωμών. Ας διορθώσουμε λοιπόν τα προβλήματα και ας αποκαταστήσουμε ένα προϋπολογισμό πραγματικά ευρωπαϊκό. Ο κύριος Σοντή θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια συμφωνία γιατί αλλιώς θα γελιοποιηθούμε στην διεθνή κοινότητα σε αυτό που έχει απομείνει σε έναν μικρό προϋπολογισμό. Η συμφωνία αυτή είναι δύσκολη όμως. Πρέπει να υπάρξει ρήτρα αναθεώρησης το 2017. Μέχρι το 2017 τα κράτη-μέλη θα έχουν την δυνατότητα να επικυρώσουν το σύμφωνο σταθερότητας, θα έχουν λυθεί τα δημοσιονομικά προβλήματα και το θέμα του δημοσίου χρέους. Το 2017 θα έχουμε ένα νέο κοινοβούλιο, μια νέα επιτροπή και ένα νέο πρόεδρο του Συμβουλίου. Γι' αυτό λοιπόν ας ξεκινήσουμε με πολιτικό τρόπο να συζητήσουμε τα θέματα αυτά και ας εμείνουμε σαν Κοινοβούλιο στην ρήτρα αναθεώρησης που θα επιτρέψει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ορίσει πολιτικές και προοπτικές που να αξίζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Μάνκα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε σε κάποια κράτη δεν θα γίνει καμία δημόσια επένδυση χωρίς το Ταμείο Συνεχής και χωρίς δημόσιες επενδύσεις θα, έρθει θα βρεθεί σε τέλμα η οικονομία. Η πολιτική συνοχής φέρνει πολλά πλέον όχι μόνο στα φτωχότερα κράτη-μέλη, αλλά λόγω ενιαία αγοράς προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα και στα πιο εύπορα κράτη-μέλη που προσφέρουν αυτό το νόχα, την τεχνογνωσία, τις υπηρεσίες. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να φανεί ε, και έχουμε και μια κοινή δήλωση των 15 κρατών μελών και των φίλων της συνοχής που υπογράφηκε στην Σλάβα στις 15 Σεπτεμβρίου τρέχοντος. Οι συμμετέχοντες είπαν πως η πολιτική συνοχής αποτελεί ένα ε, επενδυτικό μέσο κλειδί και αν εκεί μειωθεί η χρηματοδότηση δεν θα πετύχουμε τις φιλοδοξίες και τους στόχους που έχουμε στα πρόσφατα συμπεράσματα του Συμβουλίου, ούτε τους στόχους της Ατζέντα 2020. Οι συμμετέχοντες μας είπαν πως δεν υπάρχει περιθώριο μείωσης των κονδυλίων του Ταμείου Συνοχής και πιστεύω πως αυτό θα πρέπει να ληφθεί όντως υπόψη. Η κυρία Μαζέκοβιτς. Σας ευχαριστώ απέναντι μπροστά σε αυτό το δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 θα πρέπει να λάβουμε υπόψη κυρίως ότι είναι θεμελιώδους σημασία να ληφθούν οι αποφάσεις γοργά. Γιατί, διότι ζούμε σε μια περίοδο έκτηλης κρίσης και διαρωτόμαστε τι θα κάνουμε και πού θα επενδύσουμε. Και αυτό το δημοσιονομικό πλαίσιο ακριβώς μας δίνει μια ακριβή απάντηση. Πέρα από το ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε θα το κάνουμε με τη συνείδηση ότι η Ευρώπη είναι ενιαία και αδιέρετη όσον αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη και στα αστικά κέντρα και στην περιφέρεια. Γι' αυτό σε σχέση με αυτά τα θέματα δεδομένη της σύνοχή πρέπει να συνεχίσουμε με την θετική τάση του παρελθόντος. Ευχαριστώ. Σιμπάνσκι παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Συμβούλιο, Επιτροπή θα ήθελα να κάνω λόγο για την σπουδαιότητα των αθλημάτων και για το ότι στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο θα ήταν πολύ σημαντικό να είχαμε περισσότερα κονδύλια ακριβώς για για το θέμα του αθλητισμού. Υπάρχει μια πρόταση από πλευρά μας, ε, μια τροπολογία και ελπίζουμε ότι η Ολομέλεια θα την υποστηρίξει. Ο αθλητισμός διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα όσον αφορά την ανάκαμψη, ιδιαίτερα όσον αφορά και την υγεία που την προάγει και την διασφαλίζει. Θα ήθελα και να αντιδράσω από την άλλη πλευρά για την ιδιαίτερη κατάσταση στην Ουγγαρία θα ήταν δίκαιο και σωστό να μπορούσαμε να συνεννοηθούμε και να διασφαλίσουμε τα θέματα αυτά, να εξηγηθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο τι χρειάζεται η Ουγγαρία για να σημειώσει περαιτέρω πρόοδο. Το 2011 κλείσαμε με το μεγαλύτερο πλεόνασμα όσον αφορά τον προϋπολογισμό. Παρ' όλα αυτά όμως η διαδικασία ε, προσφυγής έναντι της Ουγγαρίας ε, δεν έχει αποσυρθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, η συζήτηση καταδεικνύει σαφώς ότι η πλειοψηφία των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι υπέρ ενό προπολογισμού που θα δικαιώνει του στόχου και θα μπορεί να αρθεί στο ύψο ε, των προκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Όλοι γνωρίζουμε ότι, ότι διανύουμε περίοδο κρίσης και ότι υπάρχει ανάγκη ε, λιτότητας. Όταν όμως θέλουμε από την άλλη πλευρά να πείσουμε τους ψηφοφόρους μας ε, και να υπάρχει μια υποστήριξη όσον αφορά ε, τάση περικοπών αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Πρώτον, οι στόχοι δεν μπορούν να υλοποιηθούν, αλλά πέρα και από αυτό θα αντιμετωπίσουμε δημοσιονομικές δυσχέρειες. Θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει σε βάθος τον προϋπολογισμό πώς έχει και να λάβει υπόψη ότι έτσι δεν μπορούν να υλοποιηθούν οι στόχοι μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Έχουμε διάφορα θέματα που πρέπει να συζητήσουμε στα πλαίσια του πλαισίου αυτού, γιατί θα πρέπει εδώ να ε, απηχηθούν όλες οι προτεραιότητες της στρατηγικής για το 2020 και να ανταποκριθούμε και στις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών. Θα πρέπει λοιπόν ο προπολογισμό σίγουρα να βασίζεται σε σωστά επιχειρήματα που θα προωθήσουν την ανάπτυξη, γιατί η οικονομική κρίση θα πρέπει να ξεπεραστεί το συντομότερο δυνατόν και θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη οικονομική ε, οικονομική άνθηση στην Ευρώπη, περισσότερε θέσει εργασία, να ενισχύσουμε τη θέση μα στην παγκόσμια αγορά. Όλα αυτά τα μέτρα λοιπόν χρειάζονται χρηματοδότηση, χρειάζονται πόρου και δεν θα πρέπει τα χρήματα αυτά να μειωθούν σε σχέση με την τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Αντίθετα, η πολιτική συνοχή θα πρέπει να χρηματοδοτείται περισσότερο γιατί θα επενδύσουμε σε περιοχές με προστιθέμενη αξία. Και αυτά θα ήθελα να πω στον Επίτροπο. Ωραία λοιπόν, τελειώσαμε. Μπορώ να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Επίτροπο για να απαντήσει στο όσο Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, συνάδελφε, σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας δεν θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε ένα πλαίσιο δημοσιονομικών προοπτικών χωρίς τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει λοιπόν εσείς να μας βοηθήσετε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις εξαιρετικές συνθήκες στην Ευρώπη σήμερα. Γιατί νομίζω θα πρέπει να αποδείξουμε πως γίνεται πραγματική διοργανική συνεργασία κάθε θεσμικό όργανο έχει κάποιο ρόλο να παίξει και εδώ θα ήθελα να συμπεριλάβω και τα εθνικά κοινοβούλια για το θέμα της φορολογίας και των ίδιων πόρων όχι φορολόγηση χωρίς ε, εκπροσώπηση. Και αυτή είναι η απάντησή μου στον κύριο Χάρτοκ, ο οποίος πολύ συχνά κάνει τέτοιου είδους σχόλια και μετά φεύγει και δεν ακούει την απάντησή μου. Νομίζω λοιπόν πως ε, ε, αυτό ήταν ένα ε, ε, θαυμάσιο επίτευγμα το οποίο από την Ανατολική Ευρώπη εγώ θαύμαζα τα χρόνια που ήμασταν διαιρεμένοι. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να πετύχουμε και τους στόχους της ανταγωνιστικότητας για την Ευρώπη. Το κατά πόσο θα παραμείνουμε σε πολιτικές δηλώσεις ή αν θα περκοδοτήσουμε αυτή την ατζέντα με τα απαραίτητα κονδύλια. Θα πρέπει ο προπολογισμό να δει τι θα, σε τι θα επενδύσει σε πολιετές πλαίσιο στην Ευρώπη όπου δεν υπάρχουν επενδυτικά κεφάλαια στους εθνικούς προϋπολογισμούς και να δούμε ποιο θα είναι το σωστό επίπεδο, του, το ύψος του προϋπολογισμού που εδώ είναι σημαντικός ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε μια τεχνική ενημέρωση που έγινε για την συνοχή που ε, έλαβε υπόψη κάποια στοιχεία, μάλλον ατυχή, αλλά δεν μπορούμε ε, να αλλάξουμε ε, την μεθοδολογία του Βερολίνου γιατί ε, τα στοιχεία που έχουμε γιατί τα στοιχεία που χρειαστήκαμε να χρησιμοποιήσουμε θα αποτελέσουν τη μόνη η βάση υπολογισμών, αλλά θα δώσουμε κάποια χέγγια σε ε, χώρες όπως η Ουγγαρία που αντιμετωπίζουν ε, προβλήματα σε πιο πρόσφατα έτη. Για τους ίδιους πόρους το μήνυμά σας έχει να κάνει με τον τρόπο που θα χρηματοδοτηθεί ο ενιαίος προϋπολογισμός. Τι σημαίνει όμως ενιαίος προϋπολογισμός? Ε, να μην υπάρχει δεύτερος προϋπολογισμός για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ε, ενότητα συμπληρωματικής ε, φύσης ε, για τις δαπάνες και για τα έσοδα. Γιατί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το, ο, η πρόταση που έχουμε είναι ένας απλός δίκαιος προϋπολογισμός που θα ανταποκριθεί σε όσους μας ζητάνε ένα διάφανο σύστημα, δίκαιο σύστημα για τους ίδιους πόρους. Εάν λοιπόν εμείς καταφέρουμε να το παρουσιάσουμε και να μεταρρυθμίσουμε τα έσοδα, τότε θα πρέπει να κερδίσουμε και πάλι το βραβείο Νόμπελ για τις προσπάθειές μας αυτές. Τα 28 κράτη-μέλη λοιπόν ζητούν κάτι τέτοιο από εμάς. Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ένα σημαντικό ρόλο να παίξει και στις δαπάνες. Η πρότασή μας είναι μετρημένη και οι συγκρίσεις με τους εθνικούς προϋπολογισμούς είναι άδικες. Δεν υπάρχει κανένα κράτος μέλος μένα το οποίο στο παρελθόν να έχει χρειαστεί να λάβει ε, υπόψη του τέτοια διεύρυνση γεωγραφική. Θα είμαστε 28 και όχι 27 την ε, επόμενη περίοδο. Έχουμε περισσότερες αρμοδιότητες, περισσότερες ευθύνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα λοιπόν δεν μπορώ ε, να αντισταθώ στο να κάνω κάποιες συγκρίσεις. Ναι, ο ετήσιος προϋπολογισμός είναι χαμηλότερους από τον ετήσιο προϋπολογισμό από τα, από τα ετήσια ελλείμματα κάποιων κρατών μελών. Όμως, θα πρέπει εδώ να σας απαντήσω πως η συνεισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό είναι αντίστοιχο με τα όσα πληρώνει στην ε, πυροσβεστική της και λιγότερο από όσα πληρώνει για να χρηματοδοτήσει το σοφρονιστικό σύστημα στο Ηνωμένο Βασίλειο και 40 φορές λιγότερο από όσα πληρώνει για να εξυπηρετήσει το βρετανικό χρέο. Αυτά έχω να σας πω ως απάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Λεβαντός και ευχαριστούμε. Θα λάβει τον λόγο τώρα ο κύριος Mr. President. Κύριε Πρόεδρε, Αγαπητά μέλη, σας ευχαριστώ για τη συζήτηση που προηγήθηκε. Κατανοώ πλήρως και το λέω αυτό σαν εφημισμό. Κάποιοι από εσάς δεν υποστηρίζουν την πρόθεση μείωσης του συνολικού μεγέθους του δημοσιονομικού πλαισίου. Σέβομαι τις απόψεις σας, υπάρχουν διαφορές γύρω από το πολιετές πλαίσιο Υπάρχουν διαφορές όπως γνωρίζετε καλά για το θέμα αυτό και ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Ελπίζω ότι θα εκτιμήσετε ότι υπάρχουν ισχυρά επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές και διαφορετικές μορφές αντιμετώπισης για τον καλύτερο δυνατό τρόπο επίτευξης των στόχων μας. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για τον τομέα των εισόδων και θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες για τη στάση μας πάρα πολύ σύντομα. Κάποια πολύ σημαντικά θεσμικά προβλήματα για τον κοινοτικό προϋπολογισμό ήρθαν στην επιφάνεια μετά από την συνάντηση του Συμβουλίου την προηγούμενη εβδομάδα. Τέθηκαν από τον κύριο Λαμασούρ, τον πρόεδρο Λαμασούρ και άλλους εκλεκτούς ομιλητές. Αν μου επιτρέψετε να κάνω κάποια μικρά σχόλια εδώ. Ιδιαίτερα γιατί σήμερα λίγο μετά θα έχουμε την δυνατότητα να συζητήσουμε τα θέματα αυτά άμεσα με τον πρόεδρο Βαν Ένα μικρό σχόλιο λοιπόν για την παρέμβαση Γένσεν. Σέβομαι τις απόψεις σας, αλλά νομίζω ότι εμείς στην πρότασή μας δεν εκφράσαμε υποστήριξη για τη μέθοδο της δίκαιης επιστροφής, το Ζουστρετούρ, και ούτε αναφερθήκαμε χαρακτηρίζοντας ε, το θέμα αυτό σαν μια ιερή αγελάδα. Θέσαμε κάποια θέματα για αξιολόγηση. Ίσως όμως να μην κατανόησα πλήρως το περιεχόμενο της παρέμβασής σας. Για την ενισχυμένη μορφή συνεργασίας ξέρετε ότι αυτό έγινε γιατί δεν υπήρξε δυνατότητα επίτευξης του στόχου σε επίπεδο 27. Τώρα προχωράμε με την ενισχυμένη μορφή και η Προεδρία θα κάνει ό,τι μπορεί έτσι ώστε το θέμα αυτό να προωθηθεί. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όμως ότι αυτή η ενισχυμένη συνεργασία δεν αφορά ένα άγνωστος πόρος, αφορά εθνικούς πόρους. Δεν μιλάμε ε, για κάτι το οποίο είναι ένας γνωστός και χρησιμοποιούμενος πόρος. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το οποίο οποίο προσπαθούμε να κάνουμε με τον φόρο αυτό των χρηματοοικονομικών συναλλαγών από ορισμένε χώρες είναι κάτι που προσπαθούμε να συνδέσουμε με τα έσοδα των χωρών που συμμετέχουν στην συνεργασία αυτή με το θέμα των μειώσεων μέσω των συνεισφορών τους στους ιδίους πόρους. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όμως ότι εδώ υπάρχουν πολλά νομικά και πολιτικά εμπόδια σε ορισμένες χώρες εμπόδια που εμποδίζουν χώρες ε, που θα ήθελαν κατά τα άλλα να πάρουν μέρος ε, στην ενισχυμένη αυτή μορφή συνεργασίας. Θα ήθελα να υπογραμμίσω επίσης και να διαβεβαιώσω όλους όσους πήραν το λόγο μέχρι τώρα ότι οι προβλέψεις για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες είναι ένα από τα θέματα που δεν τα λίγα δυστυχώς που δεν δημιουργούν προβλήματα στα πλαίσια της συζήτηση μέχρι τώρα. Όταν λέμε εμείς ότι το επίπεδο του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου ε, θα πρέπει αναπόφευκτα να μειωθεί σε όλα τα κεφάλαια του που το συναποτελούν. Αυτό δεν είναι μια ευχή την οποία εκφράζουμε. Εμείς σαν διαιτητές, σαν διαμεσολαβητές προσπαθούμε να σας δώσουμε μία αντικειμενική παρουσίαση της ισχύουσας κατάστασης. Το ίδιο αφορά επίσης και στα θέματα του προσωπικού που έθεσε κυρίως η κυρία Ροθ Μπέρετ. Και στον συγκεκριμένο τομέα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ισορροπήσουμε λίγο τις διαφορετικές απόψεις. Να υπογραμμίσω λοιπόν για μια ακόμη φορά ότι το Συμβούλιο δεν έχει ακόμα καταλήξει σε μια θέση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Οι συζητήσεις αυτές με πραγματιστικό τρόπο συνεχίζονται με όλους όσους συμμετέχουν, με όλα τα κράτη-μέλη, το υπογραμμίζω αυτό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια εύθετη χρονικά συμβιβαστική λύση Συνεχίζουμε να εργαζόμεθα λοιπόν με τη λογική ότι τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί ακόμα ώσπου να συμφωνηθούν τα πάντα. Προχωράμε λοιπόν πολύ επιφυλακτικά, εξετάζουμε και δίδουμε την προσοχή που απαιτείται στις ενδιάμεσες εκθέσεις σας και για το ΦΠΑ και για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ακούσαμε τις απόψεις που ακούστηκαν σήμερα εδώ το πρωί και θα τις φέρουμε για εξέταση και στους συναδέλφους του Συμβουλίου. Η όσμωση ανάμεσα στις εργασίες των ε, θεσμικών οργάνων είναι ε, βασικό στόχος της Κυπριακής Προεδρίας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μαυρογιάννη. Ολοκληρώνοντας τώρα για δύο λεπτά έκαστος εισηγητές. Ξεκινάμε αλφαβητικά με τον κύριο Μπέγκε πάλι. Παρακαλώ. Παρακαλώ συνάδελφε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ πρώτα για τις παρεμβάσεις που έγιναν σε αυτή τη συζήτηση που αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό και υποστηρίζουν τις θέσεις ε, της ενδιάμεσης έκθεσής μας ε, και σε σχέση και με την ε, ψήφιση που θα διεξαρθεί. Ευχαριστώ όλους που συνεργάστηκαν για αυτό το κείμενο και θα ήθελα ευχαρίστω να πω ότι αυτή η συνεργασία με τον κύριο συνάδελφο Κάρφιν, με τους συναδέλφους της ομάδας επαφών ήταν για μένα μία από τα μία από τις πιο θετικές εμπειρίες που μπόρεσα να αποκομίσω από την θητεία μου στην Ευρωβουλή. Και αν κρατήσουμε αυτή την πορεία μέχρι τέλους θα έχουμε μια ευκαιρία κάτι να πετύχουμε χειροπιαστό και αξιόλογο για την Κυπριακή Προεδρία. Ο Προεδρεύων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με ένα νέο box για την διαπραγμάτευση όπως είπε ο κύριος Μαυρογιάννης με ένα νέο εύρος range of figures τότε μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα νέο πλαίσιο. Θα ήθελα ρητά να πω σε σχέση με την ψήφιση αυτής της ενδιάμεσης έκθεσης από σήμερα μέχρι τις 22 Νοεμβρίου είμαστε πρόθυμοι να διαπραγματευτούμε όλα τα θέματα και όλες τις λεπτομέρειες που είναι αναγκαίο να συζητηθούν ώστε να βρούμε κοινέ λύσεις για έναν αποδεκτό συμβιβασμό. Είναι δουλειά της Προεδρίας τώρα να δραθεί της ευκαιρία ώστε να μπορέσουν όλα αυτά να ενταχθούν στα τελικά συμπεράσματα και στους προβληματισμούς του Συμβουλίου 23 νοεμβριου Διότι στο τέλος τέλος και αυτό πρέπει να το ξανατονίσουμε, τα αποτελέσματα ή οι συμφωνίε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε σχέση με μια πολιτική συμφωνία δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια πολιτική εντόλη ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν και να επιτευχθεί συμφωνία στο τέλος. Διότι πρώτα απ' όλα πρέπει να εγκρίνει το Κοινοβούλιο με πλειοψηφία των μελών του ώστε να μπορέσει στη συνέχεια ομόφωνα να αποφασίσει το Συμβούλιο. Αυτό δεν θα πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε σε αυτή την αλληλουχία. Ευχαριστώ ευχαριστώ. Ο κύριος Κάλφιν έχει τώρα τον λόγο uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τη συζήτηση που προηγήθηκε. Με τη συζήτηση αυτή και ελπίζω και με το αποτέλεσμα της φοφορίας λίγο αργότερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς το Συμβούλιο. Είμαι βέβαιος ότι η Προεδρία θα μεταφέρει το σωστό μήνυμα προς το Συμβούλιο. Επίσης, Υπάρχουν τρία βασικά θέματα πάνω στα οποία θα πρέπει να σταθούμε. Από τη συζήτηση 7 βγήκαν. Πρώτον, ο προπολογισμό θα πρέπει να είναι επαρκή. Κάθε μείωση του προπολογισμού θα είναι πάρα πολύ δύσκολα αποδεκτή. Έχουμε πει επανειλημμένα ότι δεν δεχόμαστε εμείς ένα τέτοιο haircut. Δεύτερον, θα πρέπει να είναι σωστά στοχευμένος ο προϋπολογισμός και κάθε ιδέα για σωστότερη στόχευση του προϋπολογισμού θα τη συζητήσουμε, την περιμένουμε και <clears throat> αυτό χρειάζεται για να καλύψουμε τους στόχους. Και τρίτον, ο προπολογισμό αυτός θα πρέπει να βοηθά τα κρατημέλη να κάνουν πράγματα τα οποία δεν μπορούν να κάνουν αυστηρά μέσω του εθνικού τους προϋπολογισμού. Έτσι θα δημιουργήσουμε ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης, γιατί όλοι οι φορολογούμενοι έχουν κάθε συμφέρον να συμβεί αυτό. Αυτά είναι τα μηνύματα λοιπόν τα οποία θέλω να αποστείλουμε προς το Συμβούλιο. Είναι μηνύματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν κατανοητά πριν πάρει τις τελικές του αποφάσεις. Και τέλος θα επιμείνουμε στην δυνατότητα διαπραγμάτευσης όλων των μέσων που περιλαμβάνονται στις νομικές βάσεις. Ανεξαρτήτως των αποφάσεων του Συμβουλίου αυτό είναι κάτι το οποίο θα ληφθεί υπόψη και είναι κάτι το οποίο δεν θα εγκαταλείψουμε σαν δικαίωμα συμμετοχής για τους ιδίους πόρους. Άκουσα με ικανοποίηση από τον Επίτροπο Λεμαντοφσκή ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προχωρήσει με τις διαδικασίες για την ενισχυμένη συνεργασία για τον φόρο χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να μειώσουν τις συνεισφορές τους επί τη βάση του ΑΠΕΠ. Εμεί θέλουμε έναν ισχυρό και σταθερό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και θα δώσουμε μάχη γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Κάρφιν. Ολοκληρώνοντας θα λάβει τον λόγο ο πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμών, κ. Λαμασού. Ευχαριστώ πολύ. Όσο πιο δύσκολη είναι μια διαπραγμάτευση, τόσο πιο πολλοί μαζεύονται γύρω από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων και πιο πολύ αισθάνεται κανείς την πίεση να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις για, για να επιτύχει ε, το σκοπό για τον οποίο έχει βρεθεί στο τραπέζι. Θα πρέπει να δούμε τι σημαίνει η προηγούμενη συμφωνία. Μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε με την προηγούμενη συμφωνία, δεν θα χάσει κανείς, δεν θα κερδίσει κανείς, όλοι θα κρατήσουν ένα κομμάτι της πίτας και έτσι κάναμε την τελευταία φορά. Δηλαδή παρόλες τις προσπάθειες ε, του κύριου Μπάγκε και του άλλου εισηγητή τότε, κάναμε ακριβώς αυτό. Σήμερα η Κυπριακή Προεδρία έχει παρουσιάσει ένα έγγραφο για τα έσοδα του προϋπολογισμού και αναφέρεται στη συμφωνία του Φοντενεμπλό που έκανε το 84 το Συμβούλιο, δηλαδή πριν από 28 χρόνια. Τότε δεν υπήρχε καν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κύπρος η Πολωνία δεν ήταν τμήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οικονομική ε, κοινότητα ήταν 10 κράτη ε, του δυτικού κόσμου. Στην Κίνα είχαμε φτώχεια και πείνα και η ιδέα ενός ενιαίου νομίσματος ε, αναφερόταν μόνο σε κάποιες συναντήσεις σοφών. Άλλαξε ο αιώνας, άλλαξε ο κόσμος, άλλαξε η Ευρώπη τέσσερις συνεχείς διαδοχικές ε, συμφωνίες που αλλάζουν τις αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τριπλασιάστηκε ο αριθμός μελών. Όλα άλλαξαν. Και δεν άλλαξε το δημοσιονομικό πλαίσιο. Η ευθύνη μας είναι ιστορική. Η δική μας γενιά ε, αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, υπουργών, ευρωβουλευτών, ε, επιτρόπων εάν δεν πρικοδοτήσει ε, την Ευρώπη του 2020 με τον κατάλληλο προϋπολογισμό, θα μείνει στην ιστορία ε, για τις ελλείψεις της. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Λαμάσου. Η κοινή συζήτηση ολοκληρώθηκε. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα στις 12.30. Θα διακόψουμε για ένα λεπτό, ώστε να μπορέσουν να, καθίσουν οι κυρίες και κύριοι.